για την απόφαση που έχει ληφθεί για το πακέτο εταιρικών φόρων. first. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στον Επίτροπο Μοσκοβισή. To open the debate. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είχα αναλάβει την υποχρέωση εδώ και αρκετό καιρό σε μια προηγούμενη συνάντηση να σας μεταφέρω σύντομα σχετικά βέβαια κάποιες απαντήσεις στην πρόκληση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Και γι' αυτό λοιπόν τώρα πια έρχομαι εδώ για να σας δώσω κάποιες απαντήσεις επί τη βάση και των μέτρων που πήραμε πέρυσι, το πακέτο του Μαρτίου και του Ιουνίου. Υπάρχει τρόπος να δράσει κανείς το θέμα της φορολογίας των επιχειρήσεων με ξεκάθαρο τρόπο. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Στηρίξατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πολύτιμο τρόπο έτσι ώστε να έχουμε μια φορολογία δικαιότερη, διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη και σε επίπεδο περιεχομένου αλλά και σε επίπεδο πολιτικής βαρύτητας και όθησης. Δεν θα είχαμε μπορέσει να προχωρήσουμε χωρίς τη δική σας εμπλοκή. Ξέρετε ότι πολλές φορές η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συνδυάζονται, συνεργάζονται, κάτι το οποίο ε, καθιστά ε, ικανά τα μέσα αντιμετώπισης των καταχρηστικών φορολογικών ρυθμίσεων. Τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στις διάφορες εκθέσεις τις οποίες παρουσιάσατε εσείς τον προηγούμενο χρόνο από τις Επιτροπές ΕΚΟΝ και ΤΑΞ δείχνουν τις συνέργειες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μπορέσετε να διαπιστώσετε ότι και οι συστάσεις σας γίνονται εν πολλής δέκτες. Συνεπώς χαίρομαι που είμαι μαζί σας σήμερα και εκ των προτέρων θα έλεγα συμφωνούμε. Καταρχάς ξεκινάμε από μια διαπίστωση πάρα πολύ απλή αλλά και ιδιαίτερα αρνητική. Κάποιες επιχειρήσεις σήμερα δεν πληρώνουν το σωστό φόρο ή δεν πληρώνουν και καθόλου φόρο και αυτή είναι μια κατάσταση η οποία για πολλούς από τους συμπολίτε μας είναι απαράδεκτη, ανυπόφορη. Αυτή η στρατηγική θα έλεγα εποφελείται από ένα διεθνές φορολογικό και ευρωπαϊκό σύστημα που δεν είναι προσαρμοσμένο στην παγκόσμια οικονομία, μια κινητική και περίπλοκη οικονομία. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση, το πακέτο που παρουσιάζω βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Καταρχάς, μια επιβολή πραγματική και όχι θεωρητική των επιχειρήσεων. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους εκεί όπου βγάζουν τα κέρδη τους. Δεύτερον, να υπάρξει ένα ποιοτικό άλμα για την φορολογική διαφάνεια. Τρίτον, ένας υγιής φορολογικός ανταγωνισμός και μια σωστή και ευαίσθητη διασύνδεση ανάμεσα στην εσωτερική ευρωπαϊκή διάσταση και την παγκόσμια διάσταση που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Επανέρχομαι λοιπόν. Μια ουσιαστική επιβολή φόρου. Τι εννοούμε. Εμείς κάναμε κάποιες προτάσεις για να δώσουμε εγγυήσει για την πραγματική φορολόγηση των επιχειρήσεων. Αυτό τι σημαίνει. Θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή διασύνδεση ανάμεσα στην επιβολή της φορολογίας και στον τόπο όπου γεννάται το κέρδος της επιχείρησης. Και εδώ με τη δική σας στήριξη θα προχωρήσουμε με μια σύσταση και με μια οδηγία. Καταρχάς, κάναμε μια πρόταση οδηγίας την οποία θα ονόμαζα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Δεν θα πω τώρα στις λεπτομέρειες, αλλά οι πρωτοβουλίες που προτείνονται θα βοηθήσουν οι επιχειρήσεις να μην μεταφέρουν τα κέρδη τους σε σιγατρικές, σε χώρες με χαμηλή φορολογία. Και δεύτερον, όταν κάποιες επιχειρήσεις προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ρυθμίσεις αυτές, χρησιμοποιούν τα λεγόμενα υβριδικά μέσα ε, να καταπολεμήσουμε λοιπόν τις πρακτικές ορισμένων επιχειρήσεων που μεταφέρουν τα ενεργά τους, από τα ενεργητικά τους από τη μία χώρα στην άλλη για να μην πληρώνουν φόρο για αυτά. Βλέπετε ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι συμβατά με τις συστάσεις ε, των Επιτροπών ΕΚΟΝ και ΤΑΞ πέρυσι. Στην ουσία εμείς δίνουμε συνέχεια στις δικές σας προτάσεις. Η οδηγία αυτή συμπληρώνεται από μια σύσταση. Η σύσταση έχει σαν στόχο την πρόληψη της κατα... καταχρηστικής, θα έλεγα, χρήσης των φορολογικών ρυθμίσεων. Ξέρετε ότι δημιουργούνται τεχνητές διοικητικές δομές για να τύχουν ευνοϊκότερων φορολογικών μεταρρυθμίσεων μέσω συμφωνιών με τρίτες χώρες και άλλα κράτη-μέλη. Η πρότασή μας δείχνει στα κράτη-μέλη το πώς οι συμφωνίες αυτές θα γίνονται πιο, θα έλεγα, ανθεκτικές έτσι ώστε να μην υπάρχει το λεγόμενο tax shopping. Δεύτερος πυλώνας, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι η καταπολέμηση, αυτό που είπαμε ήδη, ε, των φαινομένων εναντίον της ε, διαφάνειας της φορολογικής. Θα υπάρξει και μια άλλη οδηγία λοιπόν για το λεγόμενο reporting της εκθέσεις αναχώρα αυτό το κείμενο δείχνει ότι είμαστε ε, ε, αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε τη φορολογική διαφάνεια. Τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάσουμε σήμερα το πρωί επιτρέπουν την ανταλλαγή κομβικών στοιχείων ενημερωτικών ανάμεσα στις φορολογικές διοικήσεις. Θα είμαι πιο επακριβής εδώ. Η πρόταση οδηγία θέτει σε εφαρμογή τις προτάσεις του ΩΣΑ σε σχέση με το reporting αναχώρα, με τις εκθέσεις αναχώρα θα επιτρέψουμε στις φορολογικές διοικήσεις να ελέγξουν τις μη κανονικές μεταφορές των κερδών των επιχειρήσεων. Αυτό το οποίο σας προτείνουμε σήμερα λοιπόν είναι να υιοθετήσουμε τα επίπεδα τα οποία προτείνει ο ΩΣΑ και είναι ένα πρώτο στάδιο. Γνωρίζω ότι για πολλούς από εσά αυτό δεν φτάνει. Θέλετε να προχωρήσετε ακόμα περισσότερο και να δημοσιοποιηθούν οι εκθέσεις αναεπιχείρηση. Θα ήθελα να σας απαντήσω εδώ ε, και το γνωρίζετε αυτό ότι και εγώ θα το ήθελα. Ε, το έχω πει επανειλημμένα στο εσωτερικό αυτού του σώματος και συνεχίζω να προσπαθώ σε πολιτικό επίπεδο να μην χρησιμοποιώ μια διπλή γλώσσα. Είμαι υπέρ του reporting αναχώρα ε, να δημοσιοποιείται. Απαιτείται όμως να λάβουμε υπόψη μας και κάποιες παραμέτρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μια επιμέρους πρόταση εξειδικευμένη τον Ιούνιο. Ποιο είναι το πρόβλημα. Οι υπηρεσίες μας μελετούν τον καλύτερο τρόπο τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Κάναμε μια διαβούλευση, κάναμε μελέτες επιπτώσεων και διαρωτώμεθα. Ανάμεσα σε αυτήν τη δημοσιοποίηση την οποία επιθυμείτε και εσείς όπως και εγώ, όπως και πολλοί εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την επενδυτική τους ε, δυνατότητα. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, αν όχι θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα. Ε, αυτά λοιπόν κάνουμε τώρα τις μελέτες που χρειάζεται για να μπορέσουμε να δράσουμε. Θέλουμε να είμαστε πραγματιστές και όχι απλά ιδεολόγοι γιατί η διαφάνεια και η ανταγωνιστικότητα είναι πράγματα που επιδιώκουμε από κοινού. Τρίτον, θέλουμε να αποκαταστήσουμε ένα φορολογικό ανταγωνισμό υγιή και ισότιμο ανάμεσα στις επιχειρήσεις της εσωτερικής αγοράς. Ανταγωνισμό ανάμεσα στους οικονομικούς εταίρους και ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Σε επίπεδο οικονομικών εταίρων, δηλαδή επιχειρήσεων, υπάρχει μια ανισότητα ε, στην ε, φορολογία ανάμεσα στις πολυεθνικές από τη μία και τις μικρομεσαίες από την άλλη. Τώρα γύρω με πιο συγκεκριμένους οι πολιεθνικές έχουν τα μέσα να ασκούν φορολογικές ρυθμίσεις επιθετικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνουν όλες, αλλά έχουν την δυνατότητα αυτή, διότι έχουν τεράστιες νομικές επιχειρήσεις και μια εσωτερική γεωμετρία που τους το επιτρέπει. Οι μικρομεσαίες, οι οποίες είναι ο σκληρός πυρήνας του παραγωγικού ιστού της Ευρώπης, έχουν προβλήματα, να το πούμε αλλιώς υπάρχουν σημαντικές τρευλώσεις του ανταγωνισμού εις βάρος των μικρομεσαίων που πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί. Υπολογίζουμε ότι το φορολογικό βάρος των μικρομεσαίων φτάνει το 30% περισσότερο από αντίστοιχα αυτά που πληρώνουν ανάλογα μάλλον οι πολυεθνικές. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν σαν άμεσο στόχο αυτά τα φορολογικά θέματα και ρυθμίσεις των μεγάλων επιχειρήσεων. Το πακέτο αυτό θα επιτρέψει να αποκατασταθεί μια ισότιμη και δίκαιη ανταγωνιστική κατάσταση ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε σχέση με τη φορολογική τους βάση. Ορισμένες χώρες έχουν ήδη πάρει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή και έχουν υιοθετήσει κάποιες ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν τα αρνητικά της κατάστασης. Άλλες χώρες δεν έχουν, θα είμαι ευγενικό εδώ, δεν έχουν κάνει κάτι. Είναι μια άδικη κατάσταση γιατί τα μέτρα καταπολέμησης των καταχρήσεων από ορισμένα κράτη-μέλη υπονομεύονται από πιο ε, ε, θα έλεγα φιλελεύθερες αντιλήψεις σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη. Πρέπει να υπάρξει μια ισότιμη όμως αντιμετώπιση του προβλήματος σε όλες τις χώρες μέλη. Τέλος, μια εξωτερική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρωτοβουλίες έχουν σαν στόχο να δώσουμε μια σφαιρική απάντηση σε ένα σφαιρικό πρόβλημα, να το πούμε με κάθε ειλικρίνεια. Χρειαζόμαστε μια κοινή αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπληρωματικά των εσωτερικών μέτρων τα οποία θα ληφθούν από τα κράτη-μέλη. Η νέα μας στρατηγική θα αντιμετωπιστεί επί τον κίνδυνο της φορολογικής διάβρωσης, της διάβρωσης της φορολογικής βάσης εκ των έξω καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στην Ένωση και τους διεθνείς εταίρους, ανάμεσα με τις τρίτες χώρες μάλιστα τις μη συνεργαζόμενους που συνιστούν απειλή για τη συνοχή της εσωτερικής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις χώρες αυτές για να υπάρξει μια σωστή οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό γίνεται και στα πλαίσια του G20 και στα πλαίσια του ΩΣΑ. Θα σκληρύνουμε τη θέση μας αν χρειαστεί απέναντι σε χώρες οι οποίες ακολουθούν αρνητικές κατευθύνσεις. Το πακέτο που σας παρουσιάζουμε σήμερα θα έλεγα παίρνει κάποια πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Η νέα μας ευρωπαϊκή στρατηγική προτείνει την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καταλόγου, ενός ευρωπαϊκού μητρώου των ξένων χωρών που δεν συνεργάζονται. Ευρωπαϊκού καταλόγου. Επίσης ε, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και ένα medley, ένα best of ε, των εθνικών ρυθμίσεων ε, και το τι πιστεύουν οι διάφορες χώρες μέλη για τις τρίτες χώρες, για τις έξω χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως κάτι τέτοιο δεν είναι ικανοποιητικό, αλλά παρόλα αυτά οι λίστες αυτές είχαν προκαλέσει μια συζήτηση και μετακίνησαν κάποιες χώρες οι οποίες θεώρησαν ότι φύγονται από τη συμπερίληψή τους στις λίστες αυτές και βγήκαν ήδη από τις λίστες αυτές μέσω της βελτίωσης της συμπεριφοράς τους. Τώρα η ευρωπαϊκή λίστα, όχι οι εθνικές λίστες, θα βασίζεται σε αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια τα οποία θα αποφασίσουν τα κράτη-μέλη και σε ένα συνεχή διάλογο με τις χώρες αυτές πραγματική φορολόγηση των επιχειρήσεων, φορολογική διαφάνεια, υγιής και ισότιμος φορολογικός ανταγωνισμός και εξωτερική διάσταση. Αυτοί είναι οι τέσσερις πυλώνες ε, του πακέτου καταπολέμησης της διάβρωσης της φορολογικής βάσης. Τα ε, περάσω σε μια τεχνική λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του πακέτου αυτού. Το πακέτο θα επιτρέψει να υπάρξει μια συνολική εφαρμογή των προτάσεων του ΟΣΑ. Ποιοι είναι οι παράμετροι τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει από τη μία να αποφύγουμε τις ε, διαφορετικές γεωμετρίες γιατί είναι αλήθεια ότι όλα τα κράτη-μέλη δεν είναι στο επίπεδο του όσα. Και δεύτερον να λάβουμε υπόψη μας τα ειδικά χαρακτηριστικά της εσωτερικής αγοράς. Για να αποφύγουμε μια επιμέρους εφαρμογή του BEPS της ε, διάβρωσης φορολογικής βάσης ε, και μεταφοράς κερδών απαιτείται μια κοινή αντιμετώπιση. Ορισμένες ειδικέ πρωτοβουλίες πηγαίνουν ακόμα πιο μακριά από ό,τι ρυθμίζουν τα BEPS. Ε Νομίζω ότι αυτό το κάνουμε γιατί έχουμε μάθει πολλά από τις συζητήσεις που έγιναν και εδώ μέσα και στις συζητήσεις στο Συμβούλιο. Είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε προχωρήσει σε ένα σύστημα ολοκληρωμένο και το ίδιο ισχύει σε διαφορετικό επίπεδο και στον ΩΣΑ. Είχαν τεθεί κάποια ερωτηματικά από πλευρά σα σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και την σαγίνη σε εισαγωγικά την οικονομική της Ένωσης. Να τους πω ότι οι πρωτοβουλίες που προτείνονται σήμερα το πρωί ενισχύουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι η ανταγωνιστικότητα και διαφάνεια βαδίζουν από κοινού οι προτάσεις τις οποίες θα κάνω θα αποφύγουν να υπάρξει ένας κατακαιρματισμός εθνικών ρυθμίσεων που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην εσωτερική αγορά και στις οικονομικές δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και όλα αυτά στην ουσία οδηγούν σε μια νέα φορολογική κατάσταση στην Ευρώπη υπέρ των επιχειρήσεων, αυτών που σέβονται τους κανόνες και όχι υπέρ αυτών που χρησιμοποιούν κατά το δοκούν τους κανόνες. Λίγα λόγια τώρα για να κλείσω. Καταρχά, βλέποντα μπροστά μας το τι περιμένει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι περιμένει και εσά το 16. Λοιπόν, ε, το πακέτο αυτό, ένα τμήμα του είναι ένα φιλόδοξο πακέτο, σφαιρικό πακέτο, ίσως το πιο φιλόδοξο το οποίο έχει ποτέ προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχετε ποτέ κι εσείς με τη σειρά σας εξετάσει. Δεν είναι παρά η αρχή μια σειράς πρωτοβουλειών που θα παρουσιάσουμε τους επόμενους μήνες θα έχουμε ένα άλλο μεγάλο ραντεβού σημαντικό κατά τη διάρκεια του 16. Το 16 θα είναι θα έλεγα το, της ανάκαμψης του, ε, της ρύθμισης του CCCTB στα αγγλικά. Νομίζω ότι αυτό το άξις θα μπορέσει να δώσει μια απάντηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργώντας ένα πλαίσιο ικανοποιητικό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επεξεργάζονται μία πρόταση στην παρούσα φάση, η οποία θα είναι μία πρόταση σταδιακής εφαρμογή, διότι δεν είναι δυνατόν με ένα βήμα, τουλάχιστον το Συμβούλιο δεν πίστηκε να γίνει ένα ενιαίο βήμα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να παντρέψουμε το εφικτό και το ευκταίο. Και το εφικτό περνάει από τη, σημασία, συμμαχία ανάμεσά μας, αλλά και από τη σύμφωνη γνώμη ε, των ε, κρατών μελών. Κάποιες χώρες ε, δεν έχουν πιστεί απόλυτα και γι' αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε σύμφωνα με τους κανόνες μας και να σεβαστούμε και τις κυριαρχίες των χωρών μελών. Πάντως, σταδιακά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την αφοσίωσή της στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φορολογικής απάτης. Το είπα και το επαναλαμβάνω και θα το πω για μια ακόμη φορά ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτές τις μορφές οικονομικής ανεπάρκειας που οδηγούν στην κοινωνική αδικία και ανισότητα. Οι πιο ειλικρινείς φορολογούμενοι θα πρέπει σήμερα αδίκως να υποστούν το κόστος αυτών των στρεβλώσεων. Συνεπώς λοιπόν μιλάμε για τεράστια ποσά τα οποία χάνονται. Ποσά που θα πήγαιναν στην ανάπτυξη, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νοσοκομεία, στην ασφάλεια, στα σχολεία, στις μαζικές μεταφορές και ε, στους πολίτες ε, γενικότερα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει, να εμφυσίσουμε περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη διαφάνεια και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα πρώτα μέτρα του 2015 ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Θυμίζω αυτό το οποίο γνωρίζετε καλά, η οδηγία για τα tax rulings, τις ειδικέ φορολογικές ρυθμίσεις. Έχετε προσφέρει πολλά ως προς αυτό. Το πακέτο που υιοθετούμε τώρα νομίζω είναι μια σημαντική φάση στην διαδικασία αυτή την τόσο κρίσιμη για όλους. Εύχομαι θερμότατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραμείνουν σύμμαχοι τους επόμενους μήνες έτσι ώστε η διεθνής αυτή προσπάθεια διαφάνειας της φορολογίας να γίνει ακόμα πιο δίκαιη στο μέλλον. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Λαμασούγ έχει πρώτο το λόγο στο γύρο συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα αρχικά να χαιρετήσω και το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα του πακέτου που μόλις μας παρουσιάσατε, που ενέχει σε μεγάλο βαθμό και τις συστάσεις που είχε υιοθετήσει το Κοινοβούλιο στα τέλη της περασμένης χρονιάς. Σας ευχαριστώ και για τη συνεργασία μεταξύ των θεμεσικών μας οργάνων. Ε, λυπάμαι που δεν είναι εδώ και εκπρόσωπος της Ολλανδικής Προεδρίας για να μας ε, μεταφέρει ε, τους στόχους ε, που έχει για το επόμενο εξάμεινο σε ό,τι αφορά αυτό το πακέτο. Το Κοινοβούλιο θα διδραματίσει το ρόλο του κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου για να διευρύνει το διάλογο και σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια στα κοινοβούλια των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα και όλων ε, των χωρών που ε, εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία μέσω του ΟΣΑ. Αυτό θα γίνει το Μάιο για επόμενη φορά. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπό την πίεση του, της κοινή γνώμης μετά το LuxLeaks, μια πίεση που εμείς μεταφέρουμε στα θεσμικά μας όργανα, είναι καθοδόν μια αλλαγή νοοτροπίας. Και με την υπόθεση της Google βλέπετε, για παράδειγμα, ότι για χρόνια υπήρχε μυστικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών για το ποιος θα, είναι, θα δώσει τα μεγαλύτερα κίνητρα στις μεγάλες εταιρείε για να έρθουν σε αυτή τη χώρα και τώρα βλέπουμε προσπαθούν και ανταγωνίζονται μία χώρα την άλλη για να δείξει ότι είναι αυτή που παίρνει τα περισσότερα από τις μεγάλες εταιρείε. Βλέπετε ότι είναι γελία αυτή η υπόθεση χρειάζεται εναρμόνιση της ε, φορολογική βάση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων ανά χώρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει και αυτή η αλλαγή νοοτροπία, κάποιες πολυεθνικέ θα δημοσιεύσουν ε, τα αποτελέσματά τους ε, και θα έχουν και κοινωνικές προεκτάσεις. Οι επόμενες ε, θα ακολουθήσουν. Δεν πρέπει να φτάσουν τα δικά μας θεσμικά όργανα κατόπιν εορτής. Πρέπει εμείς να ξεκινήσουμε με αυτές τις προτάσεις. Καλημέρα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Λαμασού για το ΕΛΚ. Τώρα από πλευρά ε, Σοσιαλιστών Δημοκρατών, η κυρία Φερέιρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπλήρωσε την υπόσχεσή της ε, υποβάλλοντας μια φιλόδοξη πρόταση και ακολούθησε μια οδό που συνιστά ιστορική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χειρίζεται ζητήματα άμεσης φορολόγησης. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο και ανταποκρίθηκε και, σε, και στον δημόσιο προβληματισμό όπως έχει αντικατοπτριστεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε η εταιρική φορολόγηση να οδηγεί σε αδικία μεταξύ, και άνηση μεταχείριση των επιχειρήσεων σε μια ενιαία αγορά που όλα εξαρτώνται από την δίκαιη φορολόγηση. Και υπάρχει και πίεση στα δημόσια οικονομικά. Ταυτόχρονα, να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ανταποκρίθηκε και στην πρωτοβουλία του ΟΣΑ. Όμω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταματήσει να ακολουθεί απλώ τον ΟΣΑ. Θα πρέπει να αρχίσει να ηγείται τη διαδικασία αντιμετώπιση ε, τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Και εγώ έτσι ερμηνεύω αυτές τις προτάσεις. Πρέπει να πάμε ακόμα παραπέρα. Ε, διαγράφεται η οδός και στι συστάσει του Κοινοβουλίου, το αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ευχαριστώ. Όμως υπάρχουν ακόμα ζητήματα. Για παράδειγμα, ε, τι αποτελεί φορολογικό παράδεισο. Πρέπει αυτό να προσδιοριστεί. Θα πρέπει εκεί να ενισχύσουμε τις προτάσεις μας. Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα επίση να επισημάνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προωθήσει αυτή την αλλαγή φιλοσοφία όπω ανέφερε και η Κομισιόν. Και το ξεκαθαρίσαμε αυτό και στην έκθεσή μα. Πρέπει να ενισχύσουμε το ζήτημα της, ε, ε, των συστάσεων αναχώρα, των εκθέσεων αναχώρα και να δημοσιοποιούνται και όλε αυτέ οι εκθέσει. Αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για την ενιαία οικονομία ενιαία αγορά και το ενιαίο νόμισμα. Και σε αυτό το πλαίσιο μα φαίνεται ιδιαίτερα περίεργο που δεν υπάρχει εδώ εκπρόσωπο Ολλανδική Προεδρία γιατί τα κράτη-μέλη έχουν θεμελιώδη ρόλο να διαδραματίσουν σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση τη ε, φοροαποφυγή. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τι ευθύνε του και ε, να κάνουν ό,τι μπορούν για να ενισχύσουν τη συνεργασία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω και η Προεδρία του Συμβουλίου λοιπόν να διαδραματίσει το ρόλο που τη αναλογεί. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λόνε για 1,5 λεπτό. Βρισκόμαστε στη φάση των δηλώσεων από πλευρά των πολιτικών ομάδων θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία με τις μπλε κάρτες μετά τις δηλώσεις των πολιτικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία, κύριε Επίτροπε. Ε, είναι μάλλον δυσάρεστη έκπληξη αυτές, ε, αυτή η ανακοίνωση της Επιτροπής γιατί δεν ακούμε για τις πιο αποτελεσματικές επιχειρήσεις, για το πιο αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα γιατί και οι επιχειρήσεις ε, φροντίζουν ε, για την απασχόληση. Πρέπει να υπάρχει δίκαιη μεταχείριση των επιχειρήσεων και των πολυεθνικών να μην μπορούν να φοροδιαφεύγουν και να φοροαποφεύγουν. Και πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και να μην εφησυχάζουμε. Να αγρυπνούμε σε τρία στοιχεία. Πρώτον, και για τα μικρότερα κρατημέλη, τα οποία θα πρέπει να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά του, θα πρέπει να κατέβουν ε, οι φορολογικοί συντελεστέ. Και χωρί φορολογικό, ε, χρειάζεται μάλλον και ένα υγιή φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ ε, κρατών μελών και θα ήταν κακό να υπάρξει εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, θα πρέπει να βλέπουμε και το διεθνέ πλαίσιο όταν κάποιες χώρες πηγαίνουν πέρα των όσων έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε αυτό είναι αντιπαραγωγικό για εμάς. Και τρίτον, να τηρεί το λόγο της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην υπάρχει επιπλέον άχθος ε, για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Αυτό αναφέρεται στα κείμενα της Κομισιόν. Ελπίζουμε πραγματικά να διατηρηθεί και να γίνει αυτό γιατί πρέπει να μερευνήσουμε για την μείωση τροφολογικών συντελεστών και ότι όλοι πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν. Ευχαριστώ. Από την Άλντε, Τόιρερ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δύο οδηγίες αποτελεί ένα μεγάλο ορόσημο για τη δημιουργία δίκαιου φορολογικού ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Και είναι και η πεμπτουσία αυτή των πορισμάτων της ε, Επιτροπής Τάξη που υπερψηφίστηκαν με μεγάλη πλειοψηφία εδώ στην Ολομέλεια. Γι' αυτό λοιπόν καταρχάς συγχαρητήρια κύριε Μοσκοβισή για τις προτάσεις σας ε, που συμπεριλαμβάνουν και τις ε, προτάσεις του ΟΣΑ και τι διαμορφώνουν σε ένα δεσμευτικό νομοθέτημα. Και η Άλντε είναι για την άλλη μάλλον είναι σημαντικό 28 διαφορετικές ε, χώρες να μην δημιουργούν διάφορες, ε, διάφορα παραθυράκια τα οποία εκμεταλλεύονται οι διεθνείς όμιλοι για να μειώσουν στο μετανικό συντελεστή τη φορολογία τους ουσιαστικά. Το 2014 Έξι από τις 10 μεγάλες βρετανικές επιχειρήσεις υπολογίστηκε ότι στον Εμμήνο Βασίλειο δεν πλήρωσαν καθόλου φόρο εισοδημάτων, παρά το γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο είχαν σημειώσει 30 δισεκατομμύρια λίρες κέρδη. Και είναι σαφές ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μοντέλα φοροαποφύγης, είναι σε μειονεκτική θέση. Είναι λοιπόν σαφές ότι είναι πρώτη στη ανάγκη να δημιουργήσουμε μια νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέπει ίσως όρους ανταγωνισμού. Στην Ελβετία λοιπόν και στις επισκέψεις μας είδαμε πώς μπορεί να διοργανωθεί ο ανταγωνισμός. Αυτόματο σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και κοινό ε, φορολογικό εταιρικό συντελεστή. Ε, αυτά λείπουν όμως από την πρόταση αυτή. Πότε μπορούμε να υπολογίσουμε ότι θα τα δούμε. Να δούμε τι γίνεται και στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θέλουν να ασκήσουν πίεση γιατί θεωρούν ότι θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση οι όμιλοι του. Αλλά πιστέψτε μας, θα έπρεπε να κινηθεί μαζί μας και η Αμερική προκειμένου από κοινού, Ευρώπη και Αμερική, να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε στο μέλλον σε παγκόσμιο επίπεδο τις επιθετικές μορφές φορολογήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα από την ΚΟΥΕ, ο κύριος Ντεμάζη για 1,5 λεπτό. Κύριε Μοσκοβισή, ο Σάντερς της Main Street σημείωσε σήμερα εντυπωσιακά αποτελέσματα στην πολιτεία της Άιωβα. Και αναφέρει τα, τα θέματα της ε, ε, Google και το γεγονός ότι δεν πληρώνονται φορολογία από πλευρά των μεγάλων ομίλων αυτών, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα συνεχίζουν λες και δεν έχει συμβεί τίποτα. Πρόκειται για το τρίτο πακέτο και παρόλα αυτά επαναλήφθηκε η LuxLeaks. Με τις πρακτικές αυτές ε, οι μεγάλοι όμιλοι βελτώνουν ένα 30% της φορολογησής τους και αυτό α, ξεπερνάει και τα όρια των συστάσεων του ΟΣΑ και σε ό,τι αφορά τις φορολογικούς παραδείσους. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι 5% των ε, επιχειρήσεων ε, πληρώνουν ε, τέτοιου φόρου, ενώ ο ΑΣΑ υπολογίζει το ποσοστό αυτό σε 10%. Το LuxLeaks θα έπρεπε να ονομάζεται EU Leaks, είπε ο κύριο Juncker. Έχει δίκιο. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο μαύρη λίστα για τι ποινέ και δεν μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση τέτοιων φορολογικών πρακτικών. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τέτοιες πρακτικές. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ζολή για 1,5 λεπτό από τους πράσινους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι προτάσεις τις οποίες μας παρουσιάσατε είναι ένα συμπληρωματικό βήμα για να σταματήσει η φοροδιαφυγή των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Σαν παράδειγμα, φόροι εξόδου που επιτρέπουν να φορολογηθούν άπαξ τουλάχιστον τα κέρδη που έχουν μετακινηθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς όμως οι προτάσεις είναι ατελείς και ως έχουν δεν θα θέσουν τέλος τις κοινικές φορολογικές πρακτικές. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενισχύσει το κείμενο αυτό. Δεν θέλω να ελαχιστοποιήσω την σημασία τους. Αλλά αν τα πράγματα δεν προχωρήσουν τότε η ευθύνη θα πέσει στα κράτη-μέλη που ναι μεν λένε διάφορα αλλά συνεχίζουν να ανταγωνίζονται το ένα το άλλο με καταστροφικό τρόπο. Σαν παράδειγμα αυτό που έκανε ο Όσμπορν στην Google αυτό το 3% στα 10 χρόνια είναι κάτι το οποίο στην ουσία υπονομεύει την ευρωπαϊκή συνεργασία. Κύριε Μοσχοβησή, πρέπει να δώσουμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην κοινωνία των πολιτών να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους έτσι ώστε τους επόμενους μήνες το πρόγραμμα αυτό αντιμπέψ όπως λέμε να συμπληρωθεί και οι νέοι κανόνες να γίνουν σεβαστοί και στις 28 χώρες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να στηρίξετε με ξεκάθαρο τρόπο ε, την δημοσιοποίηση των εκθέσεων αναχώρα. Η καταπολέμηση της φορολογικής αδηγίας δεν θα ολοκληρωθεί με κάποιες αποφάσεις. Δυστυχώς ο εκβιασμός στην αγορά εργασίας είναι καθεστώς. Οι υπουργοί γίνονται λόμπιστ των συμφερόντων των μεγάλων οικονομικών ομάδων. Για το EFDD έκερ, 2,5 λεπτά. Υπάρχει λόγο που θα πρέπει να αποφασίζονται οι πολιτικέ πολιτικές από τα κράτη-μέλη ε, και όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε χώρα έχει τα δυνατά της σημεία. Η Γαλλία έχει το κρασί, η Γερμανία την βιομηχανία, η Ισπανία τον τουρισμό. Αυτά δεν έχουν γίνει στερεότυπα από μόνα του. Υπάρχει λόγο. Κάθε πολιτισμό θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την ισχύ του και τη δύναμή του και στο φορολογικό του σύστημα. Ο φόρο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ε, επιλύει κάθε χώρα από μόνη τη και όχι μέσω Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η ευρωπαϊκή λύση για κάθε πρόβλημα είναι η εναρμόνιση. Ο ανταγωνισμό μεταξύ χωρών και στη φορολόγηση τη ε, παροτρύνει να έχουν και καλύτερε δημόσιε υπηρεσίε. Στην ενιαία αγορά η Google ήταν ε, ελεύθερη να πληρώσει ε, στο χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή μπορούσε να βρει. Η ευρωπαϊκή λύση δεν είναι ε, να κλείσουμε τα παραθυράκια, αλλά να ανεβάσουμε τους συντελεστές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να κλείσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να χάσουν και τη δουλειά τους χιλιάδες άνθρωποι. Δείτε τι έχει γίνει με το ΦΠΑ. Υπό το Ευρωπαϊκό Δίκαιο τα κάτι μελη πρέπει να ζητήσουν άδεια από την Κομισιόν ε, για να μειώσουν το ΦΠΑ. Όμως ε, έχουν ε, το ελεύθερο να, να ανεβάσουν το συντελεστή. Για παράδειγμα, μια ειδική φορολογική συμφωνία που έγινε για τα περιβαλλοντικά υλικά στην οικοδόμηση κτηρίων. Αυτό είναι κάτι θετικό, αλλά τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε αυτή την πράσινη συμφωνία και κατέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πάει η συμφωνία, την έκλεισαν στο σιρτάρι κάποιοι μη εκλεγμένοι δικαστές. Οποιοςδήποτε πιστεύει ότι ε, η εταιρική φορολόγηση μπορεί να διευθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν χάσει τα λογικά τους και μπορεί να χάσουν και τη δουλειά τους αν ε, υιοθετηθούν αυτές οι πολιτικές. Ευχαριστώ. Κάπελ για δύο λεπτά από το, την ομάδα ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Μοσκοβισή. Η Alphabet, η μητρική εταιρεία της Google, αυτή τη στιγμή έχει κεφαλαιοποίηση 550 δις ε, ε, η πιο ακριβή εταιρεία στον κόσμο. Ταυτόχρονα όμως ε, κατηγορείται από τις Ιταλικές Αρχές ότι φοροδιαφεύγει ε, σε ύψους 2,27 εκατομμυρίων ευρώ από τώρα μέχρι και το 2030 προβλέπεται. Και θα ζητήσει ε, και ε, επιστροφή φόρου. Αυτά προέκυψαν και από τα σκάνδαλα LuxLeaks που δημοσιοποίησαν όλα αυτά τα στοιχεία. Στο πλαίσιο της Ειδικής Επιτροπής για φορολογικά ζητήματα καθίσταται σαφές ότι 190 εκατομμύρια ευρώ χάνονται κάθε χρόνο μέσω αναποτελεσματικών φορολογικών πρακτικών και ειδικών συμφωνιών. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε, και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε την επιθετική φορολογική πολιτική και να προωθήσουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Η πρόταση της ε, Κομισιόν βασίζεται σε τρεις ε, βασικούς πυλώνες. Διασφάλιση ε, ενός αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο ήδη συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή Τάξε και θα συνεχίσει και σε ό,τι αφορά την οδηγία για την φοροαποφυγή ούτως ώστε να καταβάλλονται οι φόροι εκεί όπου παράγονται τα κέρδη. Ένα δεύτερο σημείο είναι και η διαφάνεια και εδώ θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο το Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει ε, στο θέμα αυτό της οδηγίας να προχωρήσει. Είναι σημαντικό αυτό και είναι και σημαντικό το θέμα της εκθέσης, της εκθέσης αναχώρας, αναχώρα, προκειμένου να υποχρεούνται οι χώρες μέσα σε 7 μήνες να υποβάλουν ε, τις ε, εκθέσεις αυτές. Ένα άλλο τρίτο θέμα είναι η δίκαιος ανταγωνισμός του 30% ως όριο και χρειάζεται και μια εξαιρετική διάσταση σε ό,τι αφορά τους φορολογικούς παραδείσους. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πετύχουμε ίσο ανταγωνισμό που θα ωφελήσει και τις εταιρείες. Ευχαριστώ. Από τους μη εγκεκριμένους, ο κύριος Επιτίδιος, για ένα λεπτό. Ε, ε, προκειμένου να προσελκυθούν επενδυτέ και να υπάρξει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη πρέπει να γίνεται μια ορθή και δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών στι εμπορικέ ε, επιχειρήσει. σήμερα που ζούμε στην ε, εποχή της παγκοσμιοποίησεως οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα το οικονομικό περιβάλλον και δίνουν τη δυνατότητα στις πολυεθνικές εταιρείες να παρακάμπτουν τους ε, περιορισμούς στο φορολογικό σύστημα των διαφόρων κρατών να παρουσιάζουν μικρότερα κέρδη και να κερδοσκοπούν εις βάρος των λαών όλων των χωρών. για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να υιοθετήσουμε ένα κοινό σύστημα φορολογήσεως το οποίο θα έχει ισοπεδωτικό χαρακτήρα και δεν θα λαμβάνει υπόψη του τις οικονομικές ιδιαιτερότητες των χωρών. η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια του εθνικού κράτους το οποίο κατά την εφαρμογή της δημοσιονομικής του πολιτικής μπορεί να λάβει ε, μέτρα ούτως ώστε να προστατεύσει τα συμφέροντα των μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη όχι μόνο του εθνικού αλλά και του ευρωπαϊκού συστήματος και να μην χάνουν τις ε, θέσεις εργασίας τους χιλιάδες άνθρωποι όπως δυστυχώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μου την ελλάδα. έτσι θα μπορέσει το κράτος το εθνικό να υιοθετήσει μια κοινωνική οικονομική πολιτική και κατόπιν να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα κράτη για να αποτρέψει την παράνομη και παράλογη ε, κερδοσκοπία των ε, πολυεθνικών εταιριών. Ζάλμπα Βιντεγκάιν, δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, το πακέτο το οποίο παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο Μοσκοβισή είναι κάτι το οποίο περιγράφει το πεδίο καταπολέμησης αυτής της επιθετικής φορολογικής πρακτικής των πολυεθνικών επιχειρήσεων που φύγει γενικά τα έσοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια καλή αρχή, εν πάση περιπτώσει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνονται εκατομμύρια κάθε χρόνο από φορολογικά έσοδα. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις δημόσιες παροχές υπηρεσιών, για την εκπαίδευση ή για την δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι έτοιμες να συνεργαστούν πάντα και πληρώνουν περισσότερα από κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να αποφύγουν τη φορολογία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά ακόμα και μέσω της Επιτροπής ΤΑΞ έτσι ώστε να αντιστρέψουμε την πορεία των τελευταίων χρόνων και τις ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις ανάμεσα στις πολυεθνικές και τα διάφορα κράτη-μέλη διασφαλίζοντας την διαφάνεια που είναι η προτεραιότητά μας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε εγγυήσει έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος θα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια φορολογική ε, ουσιαστική ένωση για να αποφύγουμε ένα φορολογικό ε, πόλεμο έτσι ώστε να μην υφίστανται ε, διαφοροποιήσεις ή μικρομεσαίες από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι τα σημεία τα οποία κατέθεσα από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ένα πρώτο θετικό βήμα και πρέπει να γίνουν πραγματικότητα το ταχύτερο δυνατόν. Γι' αυτό ακριβώ θα ήθελα να ζητήσω τη στήριξη του σώματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σιμών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, με ενδιαφέρον σήμερα ακούσαμε αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Μοσκοβισή. Από τη μία πλευρά έχουμε αυτούς που λένε πως οι επιχειρήσεις ε, τις έχουμε αρμέξει. Πρέπει να τις φορολογήσουμε ακόμα λιγότερο. Υπάρχουν πολυεθνικές που πληρώνουν 1% και κάτω. Δηλαδή το λιγότερο τι σημαίνει, καθόλου φόρους. Και από την άλλη πλευρά η Κομισιόν ε, λέει business as usual. Δεν τρέχει τίποτα. Έτσι πραγματικά υποτιμούμε τους εαυτούς μας. Με στην Επιτροπή Τάξε καταφέραμε να δημιουργήσουμε το κλίμα με το οποίο η Κομισιόν υπέβαλε προτάσεις που πάνε παραπέρα από όσα έγιναν τα τελευταία δέκα χρόνια. Πρέπει όλοι να πιέζουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Όλες οι επιχειρήσεις και οι πολυεθνικές να πληρώνουν δίκαιους φόρους. Να είναι διαφορετικοί από χώρα σε χώρα, αλλά δίκαιη φορολογία να πληρώνουν φόρους δηλαδή. Αυτό όμως σημαίνει πως θα πρέπει να δούμε την πρόταση της Κομισιόν και να την πιέσουμε να γίνει πιο θαραλέα και να τη στηρίξουμε. Παραδείγματος χάρη, να μην λέμε μόνο να δημοσιεύονται ποιο που πληρώνει πόσο φόρο για τις επιχειρήσεις από 57 εκατομμύρια τζίρο και πάνω, να, να κατεβάσουμε το τζίρο, το όριο, στα 40 εκατομμύρια και πάνω. Έτσι θα πιάσουμε τις περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά. Διαφάνεια λοιπόν, βασικά, βασικό αυτό. Μία έκθεση η οποία θα συγκρίνει τα πράγματα αναχώρα, επίσης θα βοηθήσει πάρα πολύ στη διαφάνεια. Εμεί θέλουμε να μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο η Κομισιόν και νομίζω πως το Κοινοβούλιο θα σας στηρίξει. Ευχαριστώ. Κύριε Βουλευτά, υπάρχει μία ερώτηση από τον ε, κύριο Ξτοφόρου. Το διέχεστε. Παρακαλώ. Πιστεύω ότι κανένα δεν αφιβάλλει ότι πρέπει να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, την φοροαπάτη, οι πολυεθνικέ επιχειρήσει να καταβάλουν του φόρου του όπω τι καταβάλουν όλε οι επιχειρήσει. Όμω εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ισοπεδώσουμε του φορολογικού συντελεστέ. Κοινό ενιαίο εταιρικό φορολογικό συντελεστή και μάλιστα ανεβάζοντα αυτόν τον φορολογικό συντελεστή, αυτό που θα πετύχουν είναι να καταστρέψουν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στι χώρε του, αλλά και οι οποιασδήποτε ξένες επιχειρήσεις θα φύγουν σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή τη στιγμή πάμε να χτυπήσουμε όσες χώρες μήνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελούν χρηματοπιστωτικά κέντρα γιατί με διαφάνεια έχουν χαμηλούς φορολογικούς συντελεστέ. Δεν φοροδιαφεύγουν, δεν κάνουν ξέπλυμα φορολογικού χρήματος, είναι με πλήρη διαφάνεια και ουσιαστικά με τον κοινό ενιαίο φορολογικό συντελεστή που αν ξεκαθαριστεί ότι δεν θα υπάρξει αλλά θα συνεχίσει ο ανταγωνισμό τότε θα προστατεύσουμε πιστεύω και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, Σα θυμίζω ότι οι ερωτήσει δεν είναι πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Απαντάτε κύριε Σίμων. Wenn Ihnen aufgefallen sein sollte, dass wir heute nicht über eine Vereinheitlichung der Körperschaft Κοιτάξτε, σήμερα δεν συζητάμε για ενιαία φορολογική βάση των ε, επιχειρήσεων. Ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να γνωρίζουμε ποια είναι η φορολογητέα ύλη επί του οποίου θα πρέπει να επιβληθεί μετά ο φόρος. Ε, το να, λέμε, το να έχουμε κατεβάσει τόσο πολύ τους φόρους ουσιαστικά στο μηδέν και πάλι να μην πληρώνονται, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κανένα αποτελέσμα. Ας, αποτελέσμα. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η φορολογητέα ύλη και μετά να εκτιμήσουμε εάν ε, και πόσο πρέπει να πληρώνουμε για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα το 1% και κάτω. Σας ευχαριστώ. Φόξ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε κυρία Μεσκοβισή. Καλωσορίζω την πρότασή σας, αλλά με επιφύλαξη. Καλό είναι ότι θέλετε νέους κανόνες για τις αποκαλύψεις για τα στοιχεία των εταιριών. Όμως οι πολυεθνικές δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες ε, στις φορολογικές αρχές και αυτό είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε τη φοροαποφυγή. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβάλει μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια και την έχει εντάξει στο επίκεντρο της ατζέντα του G8. και ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, τα μέλη ε, ξεκίνησαν αυτή την πρωτοβουλία ο ΣΑΚΕΤΖΙ 20 τη γνωστή. Όμως και εσείς συνειδητοποιείτε και καταλαβαίνετε σίγουρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί σε διεθνέ επίπεδο και όχι τόσο σε ευρωπαϊκό. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι ε, μια ακόμα δικαιολογία για περισσότερη Ευρώπη. Ε, αυτό είναι που δεν με βρίσκει σύμφωνο, γιατί είναι παρέμβαση στα δικαιώματα των κρατών μελών και δεν την επισημώ. Ε, πολιτική είναι αποκτηστική αρμοδιότητα των ε, ε, κρατών μελών. Μέσω του ΩΣΑ διασφαλίζεται ότι τα κράτη-μέλη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και παραμένουν ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι πράγματι οι πολυεθνικές θα πληρώσουν το φορολογικό μερίδιο που τους αναλογεί και ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε είναι να έχουμε ε, χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και απλούς φορολογικούς κανόνες. Ευχαριστώ. Έχετε μία ερώτηση από τον κύριο Έτεριτς. Τη δέχεστε? Έθριτς, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Φόξ. Με ενδιαφέρον παρακολούθησα το λόγο σας. Μιλάτε για ανταγωνισμό, για το επιχειρήν και φορολογικά επίπεδα για τις εταιρείες ενιαία σε ευρωπαϊκή βάση. Είναι προσωπικά για σας κόκκινη γραμμή. Και αν συνεχιστεί αυτή η κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, τι θα ψηφίζατε εσείς στο δημοψήφισμα. Εάν ένας κοινό ευρωπαϊκός εταιρικός φορολογικός συντελεστής ήταν μέρος της συμφωνίας. Απάντηση του κυρίου Φόξ. Σας ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα. Χαίρομαι διότι η φορολογική πολιτική παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και χαίρομαι διότι τα κράτη-μέλη διατηρούν το δικαίωμα της αρνησικυρίας και είμαι σίγουρος και βέβαιος ότι οποιαδήποτε συντηρητική κυβέρνηση τωρινή ή μελλοντική θα ασκήσει δικαίωμα αρνησικυρίας σε οποιαδήποτε κοινή φορολογική βάση. Άρα δεν βλέπω κάτι τέτοιο να εφαρμόζεται ποτέ. Ο κύριος Βαν Νίβενάουζεν για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα έχουμε ένα πακέτο για την φοροαποφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και την αντιμετώπιση τους. Γιατί συμφωνούμε ότι ο καθένας πρέπει να πληρώνει αυτό που του αναλογεί στους φόρους. Οι πολίτες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οπωσδήποτε και οι πολυεθνικές. Φαίνεται λοιπόν εδώ πέρα πως κάνουμε το σωστό, αλλά δεν, έχουμε ακόμα, δεν τα έχουμε ακόμα καταφέρει. Γιατί πρέπει να τα κάνουμε και σωστά τα πράγματα και βλέπουμε πως ε, δεν έχει γίνει μία μελέτη αντικτύπου. Είναι κρίμα το ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη το διεθνές πλαίσιο του ανταγωνισμού στο οποίο λειτουργούμε και είναι ευρύτατοι οι ορισμοί παραδείγματος χάρη όσον αφορά την κατάχρηση δεσπόουσας θέσης που θα οδηγήσουν οπωσδήποτε σε προσφυγές στα δικαστήρια και θα οδηγήσουν βεβαίω σε αύξηση του τζίρου των δικηγόρων αλλά κανενός άλλου. Θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε πάρα πολύ λεπτόμερος και να τα βελτιώσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, υπάρχει ένα ερώτημα για εσάς ε, κυρία Φανιούν από, από την κυρία Γραπίνη. Το δέχεστε. Κυρία Γραπίνη παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι απαραίτητο να μιλήσουμε για τις συνέπειες αυτής της ρύθμισης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υφίστανται αυτή τη στιγμή μια φορολογική πίεση τρεις φορές ισχυρότερη, βαρύτερη από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, πιστεύετε εσείς ότι με το Small Business Act υπάρχει κάτι το οποίο θα βοηθήσει ουσιαστικά τις μικρές επιχειρήσεις. Eh, ναι, κύριε Πρόεδρε, δεν ε, ξέρω αν μπορώ να το κρίνω, αλλά είναι οπωσδήποτε κρίμα το ότι στο πλαίσιο του Better Regulation Agenda του Αντιπροέδρου Τίμερμαντς δεν προβλέφθηκε αυτή η πτυχή και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έτσι νομίζω θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε τα πράγματα σαφώς ε, καλύτερα και θα μας βοηθούσε και εμάς νομίζω στις συζητήσεις μας μια καλή μελέτη αξιολόγησης του αντικτύπου. Σας ευχαριστώ για 1,5 λεπτό η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, παρά τις καλές σας προθέσεις και την καλή σας θέληση, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένει ε, πολύ στον αέρα. Δεν είναι καθόλου συγκεκριμένη. Είναι ασαφής. Και είδαμε μάλιστα χιλιάδες χιλιάδων ευρώ που χάνονται κάθε χρόνο από τους δημόσιους λογαριασμούς και ότι ε, δεν χρησιμοποιούνται εκεί που θα έπρεπε όπως το δημόσια σχολεία και αντίθετα πρόκειται για μια αύξηση φόρων ε, ε, πολύ ε, κατακόρυφη για όσους εργάζονται. Εγώ δεν έχω τίποτα κατά της κοινοποίησης αναχώρα ώστε αυτά όλα να είναι δημοσιευμένα. Ούτε έχω τίποτα εναντίον του γεγονότος ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Αλλά θέλω να ρωτήσω κύριε Πίτροπε, πότε θα αρχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα συγκεκριμένα όπου πραγματικά θα ε, αντιμετωπίζουν τις καταχρήσεις που κάνουν οι πολυεθνικές. Πότε θα μιλήσουμε σοβαρά για τον ορισμό μιας, της μόνιμης εγκατάστασης. Πότε θα ασχοληθούμε σοβαρά με τις εισαγωγές διαφόρων προϊόντων μέσω των οποίων γίνονται όλα αυτά τα σκάνδαλα. Και για να εγγυηθούμε την ε, εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών και την εμπιστοσύνη τους στο ευρωπαϊκό όραμα χρειάζονται πολύ περισσότερα. Πρέπει να αποδείξουμε ότι αξίζουμε περισσότερο από αυτές τις πολυεθνικές που συστηματικά προστατεύονται από αυτή την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Σκοτ ε, κάτω για 1,5 λεπτά. Επτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένη ότι το φορολογικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει την πραγματική επιθυμία να πλήξει ε, τη δυνατότητα των πολυεθνικών να επηρεάσουν κυβερνήσεις για να μειώσουν τη φορολογία τους. Θα πρέπει επιτέλους να τελειώσει αυτή η εποχή όπου ο λαός χυμάζεται και οι πολυεθνικές ε, είναι σε προνομιακή κατάσταση. Τώρα, ε, στο Λονδίνο οι δικοί μας ηγέτες μπορεί να κάνουν κάτι οριζοσπαστικό αλλά στις Βρυξέλλες κάνουν το παν τέτοιου, ώστε τέτοιου είδους ε, προτάσεις να μην γίνουν ποτέ νόμος. Χαίρομαι με την ε, ε καταγραφή αναχώρα, αλλά θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι Βρετανοί ηγέτες στις πρόσφατες τροπολογίες και όσο, ό, όλους όσους ψήφισαν κατά πρόσφατα για τα θέματα αυτά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μισθωτοί, όλοι αυτοί που φέρουν το φορολογικό βάρος μας, σε έχει κουράσει πάρα πολύ όλη αυτή η η ρητορική για τη φορολογία. Κάθε φορά που ξεσπάει ένα σκάνδαλο βγαίνουν οι πολιτικοί και εκφράζουν κλαφμό και οδυρμό, αλλά όταν έρχεται τώρα να ψηφίζουν, ψηφίζουν κατά ε, και ψηφίζουν ουσιαστικά υπέρ των πολιεθνικών. Όσο πράσινοι, ως μέλος της ομάδας των πρασίνων, θα παρακολουθώ στενά τη συμπεριφορά του κυρίου Όσπουρν όταν ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φτάσει στο Συμβούλιο, γιατί τότε ε, θα μπορέσουμε να δούμε αν θα μεταφράσει τα λόγια του σε πράξεις και αν θα μπορέσει ο Βρετανικός λαός πραγματικά να το συγχωρήσει και ε, να δει ότι εννοούσε αυτά που έλεγε. Τζάνι, για ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Για αυτή την πρόταση θα πρέπει να πω ότι εδώ το βουνό γέννησε ένα ποντικάκι. Ε, ε, είναι χαρακτηριστική περίπτωση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα με ακατάλληλα μέτρα. Χρειάζεται πολύ περισσότερο θάρρο, γιατί ξέρουμε ότι μετά θα πρέπει να αγωνιστούμε και κόντρα στο Συμβούλιο για να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε καλά ποια είναι η θέση ορισμένων κρατών μελών, για τα οποία μα λένε πάνω από. μα λένε πολλά λόγια. Και τώρα με την Ολλανδική Προεδρία, ε, μάλλον προσπαθεί να βρει κάποια λύση, ε, ε, να, να βρει μάλλον κάποια λύση για ένα για να προσκαλέσει περισσότερες επενδύσεις εις βάρος άλλων κρατών όπως η Ιρλανδία, το Βέλγιο ή το Λουξεμβούργο ε, του Προέδρου Γιούγκερ. Σε αυτές τις τροπιαστικές πρακτικές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λέει τίποτα γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πως δεν υπάρχει κοινή βούληση ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίθετα, ο διαγωνισμός είναι πώς θα εκμεταλλευτούμε τις διπλανές μας χώρες ε, διευκολύνοντας τις μεγάλες πολυεθνικές εις βάρος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Θα ήθελα μάλιστα να καταλάβω γιατί στην πρότασή σας δεν αναφέρει αναφέρεστε στην αναχώρα έκθεση που να δημοσιεύεται. Γιατί αυτό ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτε και αυτό αντιπροσωπεύει το μόνο τρόπο για να είναι αποτελεσματικό. Η διαφάνεια θα πρέπει να είναι το κλειδί όλων. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζουμε ακριβώς πώς ενεργούν πραγματικά οι πολυεθνικές και τα κρατημέλη. Τα, τα ίδια που λένε στα λόγια ότι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν, αλλά μετά αρνούνται να μας δώσουν τα στοιχεία, κυρώνουν όλες τις ε, ε, ε, πληροφορίες που θα μπορούσαν να τους βάλουν σε δύσκολη θέση, όπω εκβαληθεύσαμε και στην Επιτροπή Τάξη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Τζάνι. Ο κύριο Μονό, ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δύο κείμενα για την καταπολέμηση της, ε, ε των, της Συμφωνούμε με το σχέδιο Άξης και όλα αυτά τα σχέδια. Για το reporting αναχώρα είμαστε υπέρ της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων, αλλά όχι της ανταλλαγής οικονομικών στοιχείων. Ε, κάποιες από τις προτάσεις σας αποκλίνουν από τις προτάσεις του ΟΣΑ. 10% θα ήταν λογική η φοροαπαλλαγή ε, του ε, επιτοκίου πριν από το ΕΠΙΤΑ, ε, δηλαδή τα έσοδα πριν από τόκους φόρους κτλ. Τελικά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έχουν μπει στα δημόσια ταμεία. Είναι πρόοδος αυτό. Κύριε Μοσκοβισή, οι Γάλλοι επιθυμούν να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη και ελπίζω σήμερα οι φίλοι σας στη γαλλική κυβέρνηση θα πετύχουν αποτελέσματα για να ελαφρύνουν το βάρος ε, του φορολογουμένου. Ο κύριος Τίντερ Μάγερ για 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά που αποκάλυψε το Google του Ηνωμένου Βασιλείου και το LuxLeaks Αυτά τα προβλήματα δεν θα εξαφανιστούν από μόνα τους. Πρέπει να δράσουμε. Η δίκαιη φορολογία ε, δεν θα έρθει ε, εκ του μηδενός. Χρειαζόμαστε περισσότερο συντονισμό, περισσότερη συνεργασία και ε, πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε κανόνες που να... Καλωσορίζω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βασίζεται σε μια σαφή ατζέντα, που βασίζεται στο σχέδιο δράσης και τον οδικό χάρτη του ΟΣΑ και που στηρίζεται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτείνεται την εφαρμογή και υλοποίηση ορισμών βασικών συστάσεων του ΟΣΑ και έχετε τη στήριξή μου. Ελπίζω να σα στηρίξουν και οι Υπουργοί Οικονομικών στο Συμβούλιο. Είναι όμω μόνο η αρχή όλα αυτά. Πρέπει να εφαρμόσουμε όλε τι πτυχέ και να παλέψουμε γι' αυτό, να αγωνιστούμε να εφαρμοστούν όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά παντού στον κόσμο. Και υπάρχει και ένα κατάλογο ειδικών συστάσεων ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βελτίωση του κώδικα δεοντολογία, καλύτερη μέτρηση του δημοσιονομικού κενού, και ούτω καθεξής. Τέλος το CCTV σχέδιο είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχουμε καλύτερο περιβάλλον για τις εταιρείες που λειτουργούν στην Ευρώπη. Μπορείτε να βασιστείτε στη στήριξη των ε, περισσότερων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζουμε να βελτιώσετε το φορολογικό σύστημα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριος Μπαγιέ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, μετά την ελβετική υπόθεση και το LAX Leaks και την Ειδική Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσιάσατε διάφορες δέσμες μέτρων για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Είστε ο Επίτροπος με τη μεγαλύτερη φιλοδοξία να βάλει τάξη στα οικονομικά της Ευρώπης. Δεν είστε τέλειος, όμως όλες οι δράσεις σας πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να το ε, να το υποστηρίξουμε αυτό και να σας στηρίξουμε. Μετά τις συστάσεις της ειδική Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άλλοι, οι επόμενοι λοιπόν, θα είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Και θέλουμε αυτόματη και εξατλητική ανταλλαγή απόψεων ε, και πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Κάποιες συστάσεις τις έχετε αποφύγει και δεν τις έχετε περιλάβει, π.χ. να είναι δημόσιες αυτές οι ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών, δυστυχώς αλλά σε κάθε περίπτωση η δέσμη μέτρων που προτείνεται πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορεί κανείς να καταπολεμήσει έτσι τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Και η Ειδική Επιτροπή Τάξε μίλησε για την αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων και έχει και κεφάλαιο για την ενοποιημένη φορολογική βάση. Όμως, οι ζώνες κέρδους των πολυεθνικών δεν έχουν ξεκαθαριστεί με σαφήνεια ε, και αυτό πρέπει να γίνει για να πληρώσουν φόρους εκεί όπου εδρεύουν και όχι σε κάποιο φορολογικό παράδεισο όπως η Google για παράδειγμα. Το να πληρώνουν φόρους σε φορολογικούς παραδείσους είναι κάτι που πλήττει το κοινωνικό ευρωπαϊκό μοντέλο, την απασχόληση και την ασφάλεια. Το δημοσιονομικό και φορολογικό πακέτο που προτείνεται δεν έχει στόχο να εναρμονίσει το φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, γιατί αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Όμω, αν γινόταν, θα ήταν πολύ πιο δίκαιο και θα ήταν και πολύ πιο υγιέ για την οικονομία τη Ευρώπη. Ελπίζω το Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι θα σα στηρίξει και μάλιστα για να κάνετε ακόμα περισσότερα βήματα προ την κατεύθυνση που έχετε ήδη υιοθετήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λούκιο, τον οποίο δεν βλέπω, οπότε ε, τώρα το λόγο θα πάρει η κυρία Χάρκιν για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλοδεχούμενο το πακέτο αυτό. Πολλέ πολυεθνικές μέσω επιθετικού σχεδιασμού εκμεταλλεύονται παραθυράκια και ασυνέπειε στην εθνική νομοθεσία και πληρώνουν φεδρά επίπεδα φόρων που δεν έχουν ούτε μία σχέση με τα κέρδη του. Ο ΣΑ η φοροαποφυγή είναι μεταξύ 100 και 300 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τοπικό επίπεδο και 50 και 70 δισεκατομμυρίων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για χιδέα ποσά φοροαποφυγής και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Η Κομισιόν μας λέει πως η πρωτοβουλία BEPS του ΟΣΑ δεν επαρκεί, οπότε η πρόκληση είναι να προωθήσει αυτό το ζήτημα αναλαμβάνοντας ε, βεβαίως ε, ηγετικό ρόλο παγκοσμίω, ε, ενώ ταυτόχρονα δεν θα βλάψει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δρασή μας πρέπει να είναι αναλογική τέλος. Δεν είναι μόνο Συμβούλιο και Κοινοβούλιο που θα προωθήσουν το ζήτημα. Οι καταναλωτές θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό θεωρώ πως οι εκθέσεις αναχώρα θα είναι πολύ ισχυρό εργαλείο. Σας ευχαριστώ. Βιέγκας για 1,5 λεπτό. Υπόθηκε ήδη σήμερα ότι οι πολυεθνικές εταιρείες δεν πληρώνουν φόρους. Είναι αλήθεια ότι δεν πληρώνουν φόρους, όχι μόνο σήμερα, αλλά εδώ και δεκαετίες, με τη συνεργασία των κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό μέσα στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της οικονομίας και της κίνησης κεφαλαίων. Όλο ένα και πιο φανερό γίνεται ότι η πολιτική γίνεται για τους μεγάλους ομίλους. Ωστόσο, δεν μπορούμε να το αποσυνδέσουμε αυτό με, από την βαθιά φιλελεύθερη πολιτική της Ευρωπαϊκής σε Το φορολογικό πακέτο ε, είναι μια πρόταση, όμως δεν λέγεται τίποτα για την τεράστια επιρροή ε, της βιομηχανία των συμβουλατόρων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν καλό να μας πει ο κύριος Επίτροπος σε ποιον ανέθεσε την ε, μελέτη για τον αντίκτυπο στην PwC που έκανε επίσης την μελέτη για τις οικονομικέ συνήθειε των χωρών σε ποιον, γιατί 80 με 90% των πολυεθνικών εταιριών είναι ε, έχουν και τέτοιες συμβουλευτικές εταιρείε. Θα πρέπει να δούμε ότι ποιες, ποιες, ποια είναι οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από αυτές τις εταιρείε και που κερδίζουν και διαπραγματεύονται τέτοιου είδους φορολογικές απαλλαγές. Θα δούμε τα ίδια με το παρελθόν, καταλόγους με τέτοιες ε, χώρες όπως η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία ή το Βέλγιο. Πώς θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαμπέρτ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Μας έρχεστε από τη Γαλλία όλο και περισσότερο η πατρίδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αυτό πρέπει να το διαπιστώσουμε, αλλά πάντοτε είναι η χώρα της αγάπης ε, ε, και πρέπει να αναγνωρίσουμε την ε, σημασία των προκαταρτικών. Είναι αλήθεια ότι σε θέματα φορολογικής δικαιοσύνης μετά το Swiss Leaks, μετά το Offshore Leaks και το Lux Leaks τα προκαταρτικά δεν πάβουν να δεν πάβουν να τελειώνουν υποτίθεται, αλλά πρέπει να περάσουμε στην πράξη. Βέβαια μπορεί έτσι το αντικείμενο της επιθυμίας μας να φύγει. Ε, και να απογοητευτεί. Ε, Όμω τι θα πει τότε περνάμε στην πράξη. Το είπατε και εσεί ο ίδιο ε, Θα πρέπει να επιβάλλουμε αναχώρα έκθεση δημόσια και είστε υπέρ και σα πιστεύω. Πρέπει λοιπόν οι πολυεθνικέ εταιρείε να δηλώνουν πλέον όχι πια μόνο πόσο κέρδη έχουν και πόσου φόρους πληρώνουν αλλά και σε ποιο όνομα, υπό ποιο όνομα λειτουργούν, τι είδους φοροαπαλλαγές λαμβάνουν και για όλε τι χώρε και αυτό να είναι διαθέσιμο για όλους μας τους συμπολίτες. Και αυτό θα πρέπει ολοκληρωτικά να εφαρμοστεί η σύσταση του ΩΣΑ. Αλλά στο πακέτο που μας προτείνεται και που αυτή τη φορά αξίζει τον, το όνομα αυτό, ε, ότι είναι δηλαδή ένα πακέτο, ξεχνάτε κάποια πράγματα. Ας πούμε την υποχρέωση σε όλες τις διμερείς ε, συνθήκες να αναφέρονται όλα αυτά. Αυτό είναι μία σύσταση απλά. Υπάρχουν κανόνες για τις ε, υποξένο έλεγχο εταιρείε δεν αναφέρονται πλήρως αλλά πρέπει αυτό να το ξεπεράσουμε γιατί ο ΣΑ δεν ασχολήθηκε με όλα και ας πούμε αυτό το νέο όχημα το patent boxes ε, ε, τελείως ε, αγνοείται από τον ΩΣΑ το νέο εργαλείο για φοροδιαφυγή όσα ναι, κάνει προτάσεις, αλλά εσείς έχετε την πρωτοβουλία για νομοθεσία και επιτέλους θα πρέπει να υπάρχει ένα, μια κοινή φορολογική βάση για τη φορολόγηση των ε, εταιριών. Δηλαδή να συνοηθούμε τι θα πει κέρδος και αυτό να κατανοηθεί ανάλογα. Και βέβαια όλα αυτά τα αναφέρατε στην ομιλία σας ε, πάνω κάτω. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθεί η πράξη, σας πιστεύω. Αλλά εντάξει, εμπρός, ε, μην κρατιέστε άλλο, πρέπει να ξεκινήσετε. Το θέμα είναι τα κράτη-μέλη όπως ε, είπε και ο Πιέρ Μοσκοβισή, ε, έχουν, ε, διαπνέονται από φορολογική δικαιοσύνη. Αν θέλω να κρίνω από την αντίδραση του Μεγάλου Δουκάτου Λουξεμβούργου άλλων χωρών, της χώρας μου της ίδιας ή του Φέστερ Χάγκεν, πολύ αμφιβάλλω. Πριν να σβήσει λοιπόν αυτή η επιθυμία, θα πρέπει εμείς μαζί με την Κομισιόν να προκαλέσουμε ακράτητη επιθυμία, πολύ καυτή κατάσταση, για να περάσουμε επιτέλου στην πράξη, γιατί το θύματα είναι οι μικροί φορολογούμενοι, είτε είναι άτομα, είτε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μακ, ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, κατά την ε, άποψή σας ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι κάτι το κακό. Μα εγώ θεωρώ πως έτσι προστατεύεται ο φορολογούμενος από φόρους οι οποίοι ανεβαίνουν συνεχώς. Παραδείγματος χάρη στην Ελβετία το Σύνταγμα προστατεύει τον φορολογούμενο και δεν επιτρέπεται να ανέβουν στο άπειρο οι φόροι. Ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι η μοναδική δυνατότητα που έχει ο φορολογούμενος. Εσείς μιλάτε για επιθετικές φορολογικές πρακτικές, αλλά Κατά την άποψή μου, οι δικές σας οι πρακτικές είναι επιθετικές, καθώς υπονομεύεται το φορολογικό ανταγωνισμό. Κύριε Μοσκοβισή, λέτε πως έχετε επανάσταση στα φορολογικά. Δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε κάτι τέτοιο. Οι συνθήκες δεν σας δίνουν τέτοιο δικαίωμα. Δεν μπορείτε να εναρμονίσετε τους φόρους. Αναφέρεστε στο άρθρο 115 της συνθήκης. Μα αυτό είναι για την εσωτερική αγορά, όχι για τους φόρους ο στόχος σας θεωρώ είναι να πάρετε με κόλπα ένα κομμάτι των φόρων από τις χώρες για να τα βάλετε στα δικά σας ε, ταμεία. Έχω να πω το εξή ε, για τη Γαλλία. Αν σας ενοχλεί που φεύγουν οι εταιρείε λόγω των υψηλών φόρων, μειώστε τους φόρους σας και να γίνουν πιο αποτελεσματικές εταιρείε. Σας ευχαριστώ. Ροζάτη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το φαινόμενο αυτό της ε, φοροαποφυγής ε, οδηγεί στην μείωση των φορολογικών εσόδων. Είναι πηγή αθέμη του ανταγωνισμού μεταξύ εταιριών και συμφωνώ ότι προσπαθώντας να λύσουμε αυτό το πρόβλημα κατά περίπτωση σε κάθε κράτος μέλος μέχρι στιγμής δεν είχε αποτελέσματα. Γι' αυτό καλωσορίζω την πρόταση Κομισιόν για περιορισμό του φαινομένου με την υιοθέτηση μιας πρότασης ε, για μια οδηγία για τη φοροαποφυγή και μια βελτιωμένη οδηγία για την διοικητική συνεργασία. Μεγάλη σημασία εδώ πέρα έχει η οδηγία φοροαποφυγής που βασίζεται σε έξι μέσα που στόχο έχουν να καταπολεμήσουν ακριβώς την φοροαποφυγή. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη ρύθμιση όσον αφορά έναν περιορισμό μετακίνησης κεφαλαίων στο εξωτερικό και απαγόρευση Εντό των εταιριών της αποζημίωσης ε, ορισμένων θέσεων. Τέτοιε προτάσεις περιέχονται ήδη στην πρόταση BEPS του ΩΣΑ, αλλά να τονίσω πω. όλα αυτά πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις συνθήκες και ιδιαίτερα με την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Δεν πρέπει ε, να υπάρξει λοιπόν φορολογική εναρμόνιση. Επιπλέον, οι νέοι αυτοί οι κανονισμοί δεν πρέπει να επιβαρύνουν τις ε, εταιρείε μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κόφοντ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα που παρουσιάσατε αυτό το πακέτο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα στην Ευρώπη με τους τέσσερις πυλώνες. Οπωσδήποτε η φοροαποφυγή απειλεί το κοινωνικό μα κράτο. Μιλάμε για 2.000 ε, ευρώ κατά κεφαλήν ανά Αυτό μα κοστίζει η φόρο αποφυγή και η φοροδιαφυγή. Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ κοστίζει ετησίω στην κοινωνία μας. Φανταστείτε σε τι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σχολεία, εκπαίδευση, εκπαί... επένδυση στο κοινωνικό κράτος. Πλέον διακυβεύεται και κάτι σημαντικό. Όταν οι πολίτες βλέπουν πως οι πολυεθνικές πλέον σχεδόν 0% φόρους αμφισβητούν τις βασικές αρχές του κράτους. Όταν βλέπουν ότι το Βέλγιο έδωσε σε 35 πολυεθνικές εταιρείες παράνομες φορολογικές συμφωνίες, αντιλαμβάνονται πως οι πολυεθνικές είναι πιο ισχυρέ από το κράτος το ίδιο. Βλέπουν πως το φορολογικό σύστημα είναι άδικο και βλέπουν αδικία. Εταιρείε ε, και χώρες παραβιάζουν τον νόμο πρέπει να τιμωρηθούν. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο έχει διαλυθεί. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Γιατί, γιατί οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λειτουργούν στην σκιά της οικονομίας, χρησιμοποιούν τα παραθυράκια. Ως ε, εισηγητής ε, της έκθεσης για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με την Ελβετία γνωρίζω πως η διαφάνεια είναι το μέλλον και έτσι ακριβώς θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των χωρών μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν εκθέσεις αναχώρα έτσι ώστε οι πολυεθνικές να πληρώνουν τους φόρους τους και πρέπει να πληρώνουν όλοι τους φόρους τους. Λοιπόν, ελπίζω να παλέψετε όπως είπα για εκθέσεις αναχώρα για να διασφαλίσουμε την δικαιοσύνη και να προστατεύσουμε το κοινωνικό μας κράτος. Σας ευχαριστώ. Ρουόνεν Λέρνερ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η φορολόγηση των επιχειρήσεων είναι εθνική αρμοδιότητα αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί ε, μια επιθετική φορολογική πολιτική από τη φύση της ε, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τις, ε, αφορά μάλλον τις πολυεθνικές. Ελπίζω πως τα όσα είπα θα αντικατοπτριστούν και στην εργασία της Επιτροπής για την σαφές ότι ο καλύτερος συντονισμός των εθνικών φορολογικών πολιτικών είναι απαραίτητος και είναι ο μόνο τρόπος για να ε, εξαλειφθούν οι φορολογικές ανισότητες που ευνοούν τις πολυεθνικές εις βάρος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό αυτό είναι κομμάτι των συστάσεων. Ο Μάρκα Τζούκερμπεργκ έκανε πολύ θόρυβο όταν είπε ότι θα έδινε το 99% της περιουσίας του στις αγαθεργίες. Θα μπορούσε όμως να πληρώνει και κανένα φόρο μέσα σε όλη αυτή την αγαθοεργία του. Και ευχαριστώ κύριο Φέρμπερ. 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε πως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και του του φορολογικού ανταγωνισμού πρέπει να ενταθεί, αλλά θα χαιρόμουν ε, εάν το βασικό ζητούμενο εδώ πέρα ε, ήταν ε, το να εκπροσωπείται και το Συμβούλιο. Δεν είναι εδώ πέρα κανείς από το Συμβούλιο, ούτε από την Προεδρία και απογοητεύομαι πραγματικά για το ότι αυτοί οι οποίοι φταίνε εδώ πέρα αποφεύγουν και τη συζήτηση. Και κάνετε εσείς τις προτάσεις σας ως Κομισιόν που πάνε ακριβώς στη σωστή κατεύθυνση για ένα δίκαιο ανταγωνισμό ε, φορολογικό, αλλά δίκαιο, όχι αθέμητο. Γι' αυτό υποστηρίζω αυτή την ε, πρόταση και ελπίζω αυτά τα οποία συμφώνησαν τα κράτη-μέλη στο επίπεδο του ΟΣΑ, τουλάχιστον δηλαδή την πρωτοβουλία BEPS, να την, εφαρμογή, να την εφαρμόσουν και να την στηρίξουν. Και βεβαίως ε, για τις φορολογικές συνεννοήσεις με εταιρείε δεν δείχνουν καμία ιδιαίτερη όρεξη οι χώρες να αποκαλύψουν το τι συμβαίνει. Ελπίζω λοιπόν ε, να τα δει κάπως πιο σοβαρά αυτά τα πράγματα το Συμβούλιο και ενθαρρύνω την Κομισιόν να συνεργαστεί μαζί μας, να αυξήσει την πίεση στα κράτη-μέλη προς όφελος του φορολογούμενου που δεν μπορεί να ξεφύγει του μικρομεσαίου επιχειρηματία, του υπαλλήλου. Όλοι αυτοί χρειάζονται να προστατευτούν. Σας ευχαριστώ. Μορέλ για ένα λεπτό παρακαλώ. Oui, merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Επίτροπος Μοσκοβισή είπε ότι έπρεπε να ενεργήσουμε γρήγορα και, και Ξεκάθαρα και όλοι μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο και από αυτή την άποψη τα μέτρα που παρουσίασε σήμερα το πρωί είναι αναμφίβολα ένα θετικό ε, σημάδι. Ακούω του συναδέλφου που λένε επιτέλου ε, τελικά μάλλον αυτά τα μέτρα δεν είναι στο ύψο ε, τη υγιού και, και με τη ανάκτηση των Ευρωπαίων μετά από την αποκάλυψη τη υπόθεση LuxLeaks. Αλλά α μετρήσουμε και τι έχουμε κάνει, α εκτιμήσουμε και τι έχουμε κάνει. Υπάρχουν κάποιε προτάσει επιτάπητο που ποτέ δεν θα μπορούσε κάνει να τι φανταστεί καν πριν από μερικά χρόνια. Θα πρέπει να εντοπίσουμε και τι αντιστάσει, κύριε Λαμπέρ γιατί το πρόβλημα δεν είναι τόσο η Κομισιόν, εν πάση περιπτώσει όχι η Επίτροπος Μοσκοβισή, αλλά το Συμβούλιο που προφανώ και δεν θέλει να προχωρήσουν τα πράγματα. Και επίση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένα βήμα. Ένα βήμα μόνο και πρέπει να γίνουν πρόοδοι. Πρέπει να ξέρουμε να αγκαλιάζουμε τι ε, προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση επιχειρήσεων. επίση όσον αφορά τι αναφορέ αναχώρα ιδιαίτερα υπέρ τη διαφάνειας, γιατί ακούω του δεξιού συναδέλφου και θέλω να του πω ότι η διαφάνεια δεν είναι αντίθετη με την ανταγωνιστικότητα, Αντιθέτω μάλιστα και κυρίως σήμερα. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε φάση ε, με φάση, στάδιο προ στάδιο, γιατί ε, αυτό αφορά 10 με 15% των πολυεθνικών. Μιλώ για το εκθέσει. Και έπειτα τη δημοσίευση των εκθέσεων αναχώρα. πάντω συνάδελφοι, να αναγνωρίσουμε ότι πάμε προ τη σωστή κατεύθυνση. Ε, ε, πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρα και μπορούμε να έχουμε μια καρποφόρα συνεργασία με το Συμβούλιο. Αυτό που μετράει είναι και η σχέση δυνάμεων με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μόρελ, έχετε μια μπλε κάρτα. Ο κύριος Λάμπερτ, μάλιστα. Ναι κύριε Μόρελ, επειδή με αναφέρατε και μου απευθυνθήκατε σε μένα, δεν θα ήθελα να, να παρεξηγήσετε τα όσα είπα. Όσαν είπα ότι τα προκατακτικά είναι σημαντικά, είπα ότι έχουν ουσία. Δεν είναι μόνο η πράξη η οποία έχει ουσία. Δεν αρνούμε ότι τα προκαταρτικά που ξεκίνησαν εδώ και κάποιους μήνες από την Κομισιόν έχουν ουσία. Λέω απλά και μόνο ότι κάποια φάση πρέπει να ολοκληρωθεί και η πράξη. Κύριε Μορέλ, αγαπητέ συνάδελφε Λαμπέρ, δεν είμαι βέβαιο ότι ακολουθώ την μεταφορά που χρησιμοποιείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί αυτό να μας κάνει να ξεφύγουμε λίγο από τα πράγματα. Πάντως όταν ακούμε τον κύριο Μοσκοβισή θα συμφωνείτε μαζί μου, έχουμε του ίδιου στόχου. Ε, ε, ε, ε, αυτός προσωπικά, εκείνος προσωπικά είναι υπέρ της έκθεσης ανά χώρα. Ναι, να περάσουμε στην, να ολοκληρωθεί η πράξη. Ναι, και εγώ θέλω να ολοκληρώσουμε, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, ε, ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, οι προτάσεις κομισιών γίνουν πολύ περισσότερο, πολύ παραπέρα από τα διεθνώς ε, συμφωνημένα. Περιορίζεται πάρα πολύ το δικαίωμα του φορολογικού ανταγωνισμού και το επιχειρηματικό κλίμα στην Ευρώπη πλήττεται. Η Κομισιόν ε, μιλάει για ίσους όρους ανταγωνισμού. Πάρα πολύ καλή ιδέα, αλλά δεν θα συμβεί. Αν δούμε τι γίνεται με τη φορολογία των λιμένων, όπως ε, μας είπε ο κύριος Φερστάχερ για την Ολλανδία το διαμέρισμα εννοώ των ε, κάτω χωρών. Εκεί πέρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις ε, για τα λιμάνια μας. Εν ολίγης η Κομισιόν λέει πως ε, θα υπάρξει μια φορολογική βάση κοινή για τις επιχειρήσεις. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός όσον αφορά την επιβολή ευρωπαϊκών φόρων γιατί έτσι θα εξαφανιστεί ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών. Έτσι λοιπόν θα υπάρξει ένα ευρωπαϊκό κράτος. Αυτό πλήττει την πολυμορφία μας και σας παρακαλώ να μην το κάνετε. Κάρας για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η εφαρμογή των απαιτήσεών μας κατά της φοροδιαφυγής, ε, της φοροαποφυγής, των φορολογικών αδικιών μεταξύ μικρών και μεγάλων αποκτά μια δυναμική και αυτό είναι σωστό. Οι προτάσεις με τα έξι υποχρεωτικά μέτρα που προτείνει η Κομισιόν δεν είναι μόνο εφαρμογή των αποφάσεων του ΩΣΑ αλλά πηγαίνουν ακόμη παραπέρα και είναι σωστές και αναγκαίες και εμείς τουλάχιστον τις χαιρετίζουμε. Εμείς θέλουμε οι έξι αυτές προτάσεις να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Παρά το ότι γνωρίζουμε πως πάρα πολλά πράγματα είναι ανοιχτά, θα πρέπει να υπάρξει μια πρόταση για ενοποίηση της φορολογικής βάσης των επιχειρήσεων. Ακόμα είναι ανοιχτό και εκρεμεί το εάν θα υπάρχουν προτα... εκθέσεις αναχώρα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Είναι ανοιχτό ακόμα για το εάν θα εφαρμοστεί πλήρως η οδηγία περί ΦΠΑ κύριε Λάγκη. Και ακόμα παραμένει ανοιχτό το εάν θα τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι διέπραξαν τα δικήματα... αντί να επιβραβεύονται κιόλας και να πηγαίνουν τα πρόστιμα στα ταμεία των κρατών. Έχουμε πολλά να κάνουμε, αλλά τουλάχιστον έγινε ένα σωστό πρώτο βήμα. Σας ευχαριστώ. Κοφεράτη για 1,5 λεπτό. Σέρτζο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, το λέω με κάθε ειλικρίνεια ότι οι γραμμές που περιλαμβάνονται στο πακέτο το οποίο μας ε, περιγράψατε μας βρίσκουν ε, σύμφωνους, αλλά το περιεχόμενο του πακέτου όχι. Δεν είναι σύμμορφο προς αυτές τις γραμμές. Απέρο απέχουν από τις απαιτήσει που εσείς ε, παρουσιάσατε, δηλαδή να υπάρχει μια φορολογική συμπεριφορά σεβασμού από πλευρά των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτό που λείπει ε, δεν είναι μόνο η πρόταση λεπτομερή που θα έρθει, αλλά η ιδέα ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για ορισμένα από τα πιο λεπτά ζητήματα. Ας πούμε το country by country. Ε, οι υποδείξει του ΣΑ ε, ε, εγκλωβίζουν αυτές τις ε, διατάξεις μέσα στο πλαίσιο των των εφοριών. Δεν είναι διαφανής για τους πολίτες. Αντίθετα, όμως έπρεπε εμείς να είμαστε πιο διαφανείς και καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας και είναι δίκιο ε, και σωστό να ολοκληρωθεί η πρότασή σας γύρω από τις αξιολογήσεις αντικτύπου. Το ξέρετε όμως και ο ίδιος ότι όταν έγινε αυτή η δουλειά για τις τράπεζες διαπιστώσατε ότι η διαφάνεια δεν καθιστούσε εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα Αντιθέτω, το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τι επιχειρήσει, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή και η διαφάνεια να είναι το θεμέλιο. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα. Όπω είπατε και συμφωνώ ότι η διάταξη και το πακέτο αυτό είναι βιαστικό. Άμα το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι βιαστικά, όταν θα έχετε ολοκληρώσει το πακέτο, μην κάνετε οδηγία, τοποθετήστε αυτά όλα μέσα στην οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων και θα έχουμε έτσι γλιτώσει ένα σωρό μήνες και θα είναι πιο και ουσιαστική η ιδέα της γρήγορης παρέμβασης. Ευχαριστούμε ο κύριος Χέρκμαρκ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δέσμη μέτρων. Είναι σημαντικό να έχουμε δίκαιη φορολογία για να καταπολεμήσουμε τη φοροαποφυγή. Πρέπει να είναι διαφανής επίσης ως προς τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει όμως να είναι και κάτι άλλο που τίνουμε να λησμονούμε σε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ανταγωνιστική οικονομία. Και για να είμαστε δίκαιοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο υψηλά φορολογούμενη περιοχή στην παγκόσμια οικονομία και σίγουρα δεν έχουμε και τρομερή ανάπτυξη. Ούτε την πιο καινοτόμα ανάπτυξη των επιχειρήσεων και είναι ένα από τα προβλήματα που συζητούμε εδώ αυτό. Και πρέπει αυτή την οπτική γωνία να τη λαμβάνουμε υπόψη κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής δεν θα πάνε τόσο μακριά όσο αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή προτείνει κάτι που θα πάει ακόμα παραπέρα σε σχέση με τους Αμερικανούς και αυτό θα, έχει, θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα. Σε μια ψηφιακή οικονομία δεν είναι και εύκολο, ξέρετε, να πει κανείς πού ακριβώς εκτιλήσεται η δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Αυτό ήταν εύκολο στην παλιά βιομηχανική οικονομία και βιομηχανοποιημένη οικονομία. Το σημαντικό είναι να υπάρχει εξαιρετική διαφάνεια, δίκαιο παιχνίδι και ανταγωνιστικότητα και πρέπει το Κοινοβούλιο με την Επιτροπή να συνεργαστούν ακόμη πιο στενά γιατί η Ευρώπη δεν έχει γίνει ακόμα η ανταγωνιστική οικονομία που θέλουμε να είναι. Η κυρία Γκίλ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι ιστορική στιγμή. Ή θα πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα ή θα συνεχίσουμε με το σύστημα που θεσμοθετήθηκε το 1928 και το οποίο δεν μπορεί να αντικατοπτρίσει την ψηφιακή οικονομία. Θέλουμε παιχνίδι επί ίσους, ίσους όρες, ίσους κανόνες για όλους, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ηγετικό ρόλο. Πρέπει να έχει και ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Η απουσία της Ολλανδικής Προεδρίας από τη σημερινή συζήτηση είναι εξόχως απογοητευτική. Επίτροπε, καλωσορίζω τις προτάσεις σας γιατί στηρίζουν την ανάγκη να μοιράζουν μοιραζόμαστε τα κράτη, τα στοιχεία και τις πληροφορίες ε, μεταξύ μας έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο δύσκολο για τις πολυεθνικές να αποφύγουν φορολογικές διοικήσεις αναλόγως και να κάνουν παιχνίδι και να, τελικά να πληρώνουν λιγότερους φόρους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολυεθνικές να παρακάμπτουν φορολογικές διοικήσεις. Πρέπει να κλείσουμε τα παραθυράκια και να διασφαλίσουμε ότι αυτά εφαρμόζονται με συνέπεια, με συνοχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να έχουμε με ένα κατάλογο φορολογικών παραδείσων είναι ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Σύμφωνα με τους χθεσινούς Times, τέτοιου είδους συμφωνίες όπως αυτή της Google δεν είναι ασυνήθιστες στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Άστρα Ζενέκα και η BP και η Exxon Shell τελικά δεν έχουν πληρώσει φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να έχουν παραβεί κανένα νόμο. Γι' αυτό και πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο για να υπάρχει δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες. Ευχαριστώ. Σας θυμίζω να τηρείτε το χρόνο σας γιατί ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο που είχε προβλεφθεί για τη συζήτηση. Μου Σάννα, Να μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήσασταν πολύ γενναιόδωρος με το χρόνο που μας δώσετε σήμερα το πρωί. Καλωσορίζω την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δέσμη μέτρων για την ε, εταιρική φορολογία. Την περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και καλωσορίζω την νέα ενοποιημένη φορολογική βάση, την πρόταση για αυτήν που είχε παρουσιαστεί το 2011, αλλά ε, πολύ λίγα έχουν γίνει για να εφαρμοστεί έκτοτε. Πρέπει να σημειωθεί περισσότερη πρόοδο και πιο γρήγορα. Μέχρι σήμερα οι μεγάλε πολυεθνικές έχουν εξαιρετικά φορολογικά ωφέλη ει βάρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ανοίξει το δρόμο έτσι ώστε το παιχνίδι να είναι επίσης όρης μεταξύ μικρομεσαίων και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Πρέπει να είναι το περιβάλλον πιο φιλικό για οποιαδήποτε εταιρεία δραστηριοποιείται στην ενιαία αγορά, μικρή και μεγάλη το να είναι δίκαιη η εταιρική φορολογία προστατεύει και την απασχόληση στην Ευρώπη. Επίσης, ε, το επιχειρήν, η δημιουργία startup νεοφιών και νοτόμων επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Έτσι θα έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Ε, οι επιχειρήσεις μας θα έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην Ευρώπη και πρέπει οι συνθήκες και οι προποθέσει να είναι ίσες για όλες τις ε, εταιρείε και να βελτιωθεί ο συντονισμό. Έτσι μπορεί η Ευρώπη να καλύψει την απόσταση που ε, την απόσταση που μέχρι σήμερα. Όλα αυτά θα είναι τα θεμέλια για μια πραγματικά ενοποιημένη ενιαία αγορά τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και που το χρόνο σας. Τάγκα, ένα λεπτό, παρακαλώ, Πολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, υπάρχει μια πολύ υποσχόμενη ιστορική ευκαιρία να πάψει αυτή, να καταργηθεί αυτή η βιομηχανία φοροαποφυγής η οποία δεν οδηγεί σε ισότιμο ανταγωνισμό ανάμεσα στις χώρες, όπως ίσως προτείνουν ορισμένες σε αυτή την αίθουσα. Όχι, ε, χρησιμοποιείται η ζούγκλα των εθνικών φορολογικών νομοθεσιών όπου ο δυνατότερος υπερισχύει. Δηλαδή οι μεγαλύτερες εταιρείες δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρους. Ε, καλωσορίζω αυτή την πρωτοβουλία από την Κομισιόν και εντυπωσιάζομαι από την, από την απουσία της Ολλανδικής Προεδρίας ε, και διαρωτώ με μήπως αυτή η ευκαιρία τη χρησιμοποιούμε στο maximum. Έχω δύο πράγματα να πω. Υπάρχει, ε, υπάρχει κίνητρο για κάθε τα κράτη-μέλη για να φτάσουν σε ακόμα πιο χαμηλή φορολόγηση και η ερώτησή μου είναι τι έγινε με εκείνη την ιδέα του μίνιμουμ αποτελεσματικού φορολογικού ποσοστού που προτάθηκε από κάποια κράτη και ακόμα και αν αυτή η πρόταση εμποδίσει κάποιο είδος φοροαποφυγής θα αναπτύξουν νέους τρόπους οι βιομήχανοι της φοροαποφυγής. Είναι σαφές ότι χρειάζεται αναχώρα έκθεση για να σταματήσει εντελώς αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριος Μπάλτ σε δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Από τη σκοπιά του ΕΛΚ είναι σημαντικό το ότι η Κομισιόν προσανατολίζεται στις συστάσεις του ΟΣΑ. Η Ευρώπη δεν είναι νήσος απομονωμένη. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση για να διασφαλίσουμε και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και βεβαίω δεν πρέπει να ξεχνάμε πω το θέμα δεν είναι μόνο η Ευρώπη αλλά και οι τρίτες χώρες που πρέπει να ακολουθήσουν. Έτσι θα πρέπει να βοηθήσουμε να επιτύχει η διαδικασία του όσα χαιρετίζουμε και τις περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις που προτείνει η Κομισιόν για να καταπολεμήσουμε την φόρο αποφυγή. Τώρα επιτέλους θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πράξεις και χαιρετίζουμε την πράξη σας, το ότι δηλαδή θα προσπαθήσετε να βοηθήσετε να επιτευχθεί η απαραίτητη ομοφωνία στο Συμβούλιο. Οπωσδήποτε θα δει και θα παρακολουθήσει η Επιτροπή μας και θα στηρίξει τις ε, προτάσεις σας αυτές πληροφορίες ε, βεβαίως θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για να δούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά και θεωρώ επίσης σωστό το ότι το πεδίο εφαρμογής θα επικεντρωθεί στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το να δίνουμε αναφορά για όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν δικαιολογείται. Το να δίνεται αναφορά για κάθε επιχειρήση, όπως είπα, δεν είναι και αναλογικό. Επιπλέον, θα ε, δούμε ακριβώς το τι κάνουν οι μεγάλες και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ακριβώς εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια σαφής διάκριση. Το τι κάνει η Google μας καθιστά σαφές πως πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή συνεννόηση. Γιατί όλα αυτά τα οποία βλέπουμε πραγματικά ανήκουν στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ. Χουαρέγουια για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η πλειονότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζει το σχέδιο του Επιτρόπου Μοσκοβισή. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι θέλουν να καταπολεμήσουμε τη φοροαποφυγή που οδηγεί σε οικονομική αναποτελεσματικότητα και σε κοινωνική αδικία. Όπως το είπατε πολύ σωστά, θα είναι όμως μακρά η πορεία, δύσκολη, επίπονη. Και θέλω να τονίσω δύο εμπόδια. Το πρώτο βρίσκεται εντός της ευθούσης πολλές πολιτικές ομάδες και πολλά κόμματα εντός και εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεκδικούν ε, η φορολογική αρμοδιότητα να είναι στα κράτη-μέλη, να παραμείνει και ότι αυτό είναι σωστό και καλό από την οικονομική σκοπιά. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω ότι είναι καλό πράγμα. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο σε μια ενιαία αγορά να θεωρήσουμε ότι το κάθε κράτος ενώ έχει ίδιο νόμισμα να μπορεί να έχει φορολογική αρμοδιότητα αποκλειστική για τα του οίκου του και ότι αυτό είναι υπέρ του θεμητού ανταγωνισμού και όχι του αθέμητου. Δεν το θεωρώ Σίγουρα πρέπει να υπάρχει συντονισμός για να υπάρχει ε, φορολογική διοίκηση. Αυτά τα δύο εμπόδια είναι πολύ σημαντικά κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Ρέγνερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το πακέτο αυτό τίποτε, συνεισφέρει στην φορολογική δικαιοσύνη. Η φορολογία πρέπει να ε, ισχύει για όλους, για επιχειρήσεις και για ιδιώτες. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια πορεία προς ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Η αρχή ότι οι πολυεθνικές ε, επιχειρήσεις, π.χ. τα McDonald's, ε, πρέπει να θεωρούνται μία επιχείρηση, και όχι μία λυσίδα franchise και ανεξαρτήτων καταστημάτων πρέπει να εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο όμως δεν βλέπω εγώ και ανέφεραν οι προλαλήσαντες είναι το περισσότερο θάρρος για περισσότερη διαφάνεια. Μόλις μίλησα με τον Ολλανδό πρέσβη, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι όταν ακριβώς θα έρθει η μελέτη επιπτώσεων θα ασχοληθεί το Συμβούλιο με το θέμα. Αυτό το οποίο δεν βλέπω επίσης είναι προτάσεις για την πνευματική ιδιοκτησία, τα patent boxes. Εδώ πέρα θα ήθελα λίγη περισσότερη φιλοδοξία. Ευχαριστώ Τζάνι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως μπορούμε όλοι να πούμε πως ε, το πακέτο των μέτρων που παρουσίασε η Κομισιόν πάει σωστή κατεύθυνση και ήρθε και την σωστή στιγμή. Και την συγχαίρω γιατί μπορούμε να πούμε πως προσπαθούμε όλες οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη να πληρώνουν φόρους εκεί όπου δημιουργούν τα κέρδη τους και θεωρώ πως αυτό θα συνεισφέρει και στην διαφάνεια. Η φορολογική παραδοσή εξορισμού και το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν περιέχονται σε αυτό το πακέτο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα όσο οι πολυεθνικές πληρώνουν το ένα τριακοστό των φόρων που θα έπρεπε ή αντιστρόφως αν θέλετε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληρώνουν 30 φορές περισσότερο. Φορολογούμενος στην Ευρώπη μπορεί να θεωρείται όποιος πληρώνει και μία, όσο και μία μικρομεσαία επιχειρήση. Σας ευχαριστώ. Ε, κοιτάξτε, ε, έχουμε τώρα το ΚΑΤΣΔΙ, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ σύντομοι, γιατί έχουμε προβλέψει την επίσημη πανηγυρική συνεδρίαση στις 12 με τον Πρόεδρο της Εστονίας. Ένα λεπτό λοιπόν παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το νέο πακέτο περί διαφάνειας ε, της φορολογίας είναι σημαντικό και πιο σημαντική είναι ακόμα η εφαρμογή του. Τα κατημέλη πρέπει να εναρμονίσουν τις ε, φορολογικές τους νομοθεσίες. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει τρία βασικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν εάν θέλουμε να παρεμποδίσουμε την φοροαποφυγή. Τα κρατημέλη θα πρέπει να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους, έπειτα θα πρέπει να βελτιώσουμε την απόδοση της συλλογή των φόρων και μετά την ίδια τη φορολογία. Δεν θέλουμε τα κρατημέλη να δημιουργήσουν επιπλέον ε, φόρους για τις εταιρείε που πληρώνουν δίκαιο μερίδιο φόρων. Και τέλος έχω μια ερώτηση για τον κύριο Μασκοβισή, δεδομένου ότι να αναγνωρίσατε την εισήγηση του CCTB. Θέλω να ξέρω τι μέτρα σκοπεύετε να εφαρμόσετε ώστε να ε, εισαχθεί αποτελεσματικά το CCTB αυτή τη φορά. Ένα λεπτό παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της δέσμης μέτρων για φορολόγηση των εταιριών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στόχος αυτής της απόφασης είναι το χτύπημα της φοροδιαφυγής που πλήττει πολλά κράτη μέλη της ένωσης καθώς και φορολογικών αποφάσεων τύπου tax ruling. πρωταγωνιστές βέβαια στη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή είναι οι πολυεθνικές εταιρείες με αποτέλεσμα να διαβρώνουν την εθνική φορολογική βάση. επιπλέον με την πρακτική των ενδοομιλικών συναλλαγών που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές επηρεάζονται αρνητικά οι προπολογισμοί των χωρών και πλήττεται η οικονομία τους ενώ οι πολυεθνικές γλιτώνουν δισεκατομμύρια φόρων ευρώ για την καταπολέμηση αυτών των πρακτικών βέβαια η υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών δεν αρκεί. θα πρέπει όλα τα κράτη μέλη της ένωσης να λάβουν μέτρα ώστε οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να φορολογούνται στη χώρα όπου πραγματοποιούνται τα κέρδη τους καθώς και να σταματήσουν να καταφεύγουν σε φορολογικούς παραδείσους όπως στην ολλανδία ή στο λουξεμβούργο όπου είχαμε και το σκάνδαλο το luxleaks αγαπητέ κύριε πρόεδρε της κομισιόν που είστε παρόν. ευχαριστώ. Κύριος Φλάναγκαν, παρακαλώ. Κύριε Φλάναγκαν. Χωρίς μικρόφωνο. Δεν ζήτησα εγώ το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ε, εδώ το γράφει, λέει ο Πρόεδρος. γραπίνη λοιπόν. Με συγχωρείτε. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να ασκήσουμε πολύ κριτική, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το πακέτο αυτό είναι και ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί. Τα κράτη-μέλη παίζουν εδώ πέρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η επικουρικότητα είναι σημαντική στον τομέα της φορολογίας, αλλά σημαντική είναι να καταπο... σημαντικό να καταπολεμηθεί και η αθικία στη φορολογία πρέπει να εμποδιστούν αυτές οι πρακτικές και βεβαίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αναφέρατε τους τέσσερις πυλώνες. Πρέπει να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε τα όσα λέμε. Και καλό είναι να μ' ακούει και ο κύριος Επίτροπος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ουρτασούν, φαντάζομαι ότι η Επιτροπή γνωρίζει πόσο θυμώνει ο κόσμος όταν βλέπει ότι η Κομισιόν με σιδηρό χέρι επιβάλλει λιτότητα στα κράτη, αλλά από την άλλη είναι πολύ ευέλικτη για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Σε αυτή τη δεσμή μέτρων, είναι να επιβάλλεται το πλαίσιο του G20 και μάλιστα με ντροπαλό τρόπο. Κύριε Επίτροπε, να είστε πιο φιλόδοξος, αυτό θέλουμε και αυτό χρειαζόμαστε. Να εξηγήσουν οι επιχειρήσεις αναχώρα που έχουν έσοδα και τι και πόσα, πόσα μεταφέρνουν από το ένα κράτος στο άλλο, ένα ελάχιστο συντελεστή για τις εισφορές, είναι πολύ σημαντικό η Κομισιόν να συμμαχίσει με το Κοινοβούλιο για να κάμψει τις αντιστάσεις των κρατών μελών. Για να το καταφέρουμε πρέπει εσείς να είστε πιο φιλόδοξος. Ευχαριστώ κύριος Χρυσόγονος. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της σχεδιασμένης φοροαποφυγής των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων περιέχει εύστοχες διαπιστώσεις για το μέγεθος του προβλήματος και μεγαλόστομες εξαγγελίες για την αντιμετώπιση του στο μέλλον στην πράξη όμως δεν έχει γίνει τίποτα για να διασφαλιστεί ότι ο προβλεπόμενος φόρος θα καταβάλλεται εκεί όπου παράγεται η αξία ή υπάρχει κατανάλωση. στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για δέσμη νομοθετικών προτάσεων που θα περιλαμβάνει πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής με χρονικό ορίζοντα το φθινόπωρο του. 2016. αν λάβουμε υπόψη ότι η μεταφορά της οδηγίας στα εθνικά δίκαια θα διαρκέσει άλλα δύο ή τρία χρόνια αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά συνιστούν απαράδεκτη χρονοτριβή τη στιγμή κατά την οποία τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών ισοπεδώνονται στο όνομα της δίθεν δημοσιονομικής εξυγίανσης. αν η επιτροπή εννοεί σοβαρά όσα λέει πρέπει να το αποδείξει αναλαμβάνοντας δράση τώρα και όχι στο μέλλον. Ε, Σας ευχαριστώ. Χαιρετίζω τον πρόεδρο Γιούνκερ που είναι παρόν στην αίθουσα μαζί μας και το λόγο δίνω στον Επίτροπο Μοσκοβισή για την απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ποιοτική συζήτηση. Περίπου 50 παρεμβάσεις παρακολούθησα που έθιξαν πάρα πολλά ζητήματα. Ε, διαπιστώνω, σεβόμενος βεβαίως τι ε, ευαισθησίες των ΜΕΝ και των ΔΕ, ότι υπάρχει συνένεση, ε, συμφωνείτε στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει τη δράση της για να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Ε, χαιρετίζω την παρουσία εδώ του Προέδρου Γιούγκερ και αυτή η δέσμη μέτρων μας δίνει δυνατότητα να έχουμε ένα φορολογικό σύστημα πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με όλους σας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του 21ου αιώνα και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο απασχόλησης. Τρεις είναι οι παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω. Για όσους ανησυχούν για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μην ανησυχείτε. Θέλω να σας ε, καθησυχάσω. Η φορολογική δικαιοσύνη, η διαφάνεια, η φορολογική δεν αντίκυνται στην οικονομική αποτελεσματικότητα. Είναι σήμερα παγκόσμιο το κίνημα της ε, καταπολέμησης της φοροαποφυγής. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνη της σε αυτόν τον αγώνα ε, κατά, της του, κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και άλλες πολλές χώρες έχουν δεσμευτεί να υιοθετήσουν ε, τις συστάσεις του ΩΣΑ και, το, ε, και δεσμεύτηκαν σε αυτό κατά τη σύνοδο του G20 πέρσι στην Αντάλια. Είμαι πεπισμένο αντιθέτως ότι οι δικέ μας επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν περισσότερη νομική ασφάλεια, θα έχουν λιγότερα διοικητικά βάρη και τέλη και έτσι θα υπάρχει ένας πιο ισότιμος φορολογικό ανταγωνισμός. Ό,τι είναι καλό για τη δικαιοσύνη είναι και καλό για τι επενδύσει. Είμαι πεπισμένος περί αυτού. Δεύτερη παρατήρηση. Πράγματι το, η μπάλα τώρα βρίσκεται στο γήπεδο των κρατών μελών και ε, σε ό,τι με αφορά πιστεύω στην καλή βούληση των κρατών μελών. Όχι από αφέλεια, αλλά διότι πιστεύω ότι θα ασκηθεί ισχυρή πίεση από την ε, ευρωπαϊκή και διεθνή κοινή ε, γνώμη και θα υπάρξει δέσμευση από πλευράς κρατών μελών. Είχαμε την οδηγία για την αυτόματη ανταλλαγή για τα tax rulings, για τις ειδικέ φορολογικές συμφωνίες μεταξύ κρατών και συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Δεν θα σας κρύψω ότι η ομοφωνία μεταξύ 28 κρατών μελών είναι πάντοτε ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Ωστόσο, εγώ δεσμεύομαι να δώσω αυτή τη μάχη, να κάνω τα πάντα, έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Χρειάζομαι όμως τη στήριξή σας και τη μόνιμη δική σας πολιτική πίεση, τη δική επιθυμία για μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε οι όμορφες δηλώσεις των κρατών μελών να μεταφραστούν και σε πράξεις. Βασίζομαι στην ενεργή σας στήριξη για να σημειώσουμε γρήγορη πρόοδο. Τρίτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Πολλοί παρεμβαίνοντες και προλαλήσαντες μίλησαν για το reporting αναχώρα και ε, πολλοί ζήτησαν αυτό να δημοσιεύεται. Σας είπα ποια είναι η επιθυμία μου και δεν το λέω για ρητορικού λόγους και σας είπα και ποια είναι η δική μου προσωπική άποψη, απολύτως ειλικρινής. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Ναι, στη διαφάνεια, ας πάμε μέχρι τη δημοσίευση υπό τον όρο ότι η δημοσίευση δεν θα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πραγματιστές και αυτό θα πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να πάμε σε μια ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ φορολογικών διοικήσεων, δημοσίων διοικήσεων, το επιθυμεί και ο ΩΣΑ αυτό. Θα επανέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση ε, πιο αργά μέσα στην, ε, στο τρέχον έτος. Να ολοκληρώσω όμως μιλώντας για την πολύ ενδιαφέρουσα και χαριτωμένη παρέμβαση του κυρίου Λαμπέρτς και του τρόπου με τον οποίο οι Γάλλοι προσεγγίζουν την αγάπη. Δεν θα ακολουθήσω αυτή τη σκαμπρόζικη οδό των μεταφορών, ωστόσο πράγματι τα προκαταρκτικά είναι απαραίτητα για μια επιτυχημένη ε, πράξη συνέβρεση. Και νομίζω ότι αποδεικνύεται αυτό, ε, του λόγου του αληθές φαίνεται, διότι το ποσοστό γεννήσεων στη Γαλλία είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Βέβαια, πάντοτε ο έρωτας κρύβει κινδύνους και έρωτας και πολιτική δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ε, στον έρωτα μπορεί να πρέπει να πάμε αργά, στην πολιτική όμως πρέπει να πάμε γρήγορα. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε Ολοκληρώθηκε τώρα η συζήτηση.